και την ημερησία διάταξη. Έχει τύχει ευρεία συζήτηση. Και σας προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε την προετοιμασία της ε, συνάντησης μας στην Κωνσταντινούπολη μέσα στο πλαίσιο αυτό και τότε μπορώ να περάσω στο κύριο πιάτο όπως είπα προηγουμένως τη σημερινή συνεδρίασης που περιστρέφεται από ένα θέμα γύρω από ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά γιατί έχετε πάρει και τις μαρτυρίες και τις εκθέσεις οι οποίες είναι τεκμηριωμένες και αυτό είναι και ένα από τα κύρια θέματα τα οποία για σας κυρία Όμεν Ρόιτεν είναι ένα από τα βασικά θέματα που συνάπτονται με την εκπόνηση της εκθέσεως της κυρίας Όμεν Ρόιτεν το θέμα της ελευθερίας ε, έκφρασης, το θέμα της προσωρινής κράτησης στα πλαίσια του αγώνα κατά της τρομοκρατίας που σήμερα έχει οδηγήσει σε πολλές ανησυχίες μεταξύ των κοινοβουλευτικών. Το ξέρω γιατί μου το έχετε αναφέρει πολλές φορές. Αλλά που κινητοποιεί και την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία η οποία έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συνειδητοποίησης της κοινή γνώμης σε σχέση με τις ε, πιέσεις και τις παραβιάσεις της ε, ελευθερίας έκφρασης στο πλαίσιο του αγώνα αυτού κατά της τρομοκρατίας. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω, και σίγουρα πολύ στην ε, Τουρκία συνδεδεμένη με το διαδίκτυο Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτήν την συζήτηση στο διαδίκτυο. Παρακολουθούν λοιπόν πολύ αυτήν την ε, σημερινή συνεδρίαση και θα θέλαμε να ακούσουμε τις ε, απόψεις των προσκεκλημένων μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να υποδεχθούμε τον κύριο Ακέν Αταλάη, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της τουρκικής Ένωσης για το Ποινικό Δίκαιο και ο οποίος είναι δικηγόρος δύο ατόμων που γνωρίζετε πολύ καλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Αχμέτ ε, Σίκ και του Νεδίμ Σενέρ. Τους γνωρίζουμε γιατί τους επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία ad hoc που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεκρότησε για τα θέματα αυτά με επικεφαλής τον κύριο Καρύμ, ο οποίος ε, ελπίζω θα έρθει και αυτό στη συνεδρίασή μας. Είναι λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριο ε, Ακίνα Ταλάη, ο δικηγόρο των δύο αυτών δημοσιογράφων και θα μπορέσει πιστεύω να μα παρουσιάσει ποια είναι τα τεχνικά προσκόμματα τα οποία έχουν οικοδομηθεί σε νομική βάση και επί τη βάση του ποινικού κώδικα για να εμποδίσουν την έκφραση ελευθερία μέσα στα πλαίσια του αγώνα κατά τη τρομοκρατία. Επίση έχουμε τον κύριο Αχμέτ Ινσελ που γνωρίζετε φαντάζομαι πολλέ φορέ έχει έλθει κατ' επανάληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι συγγραφέα, είναι ακαδημαϊκός, Καθηγητή, είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι πολύ γνωστή στην κοινωνία των πολιτών τη Τουρκία και είναι ένας από αυτούς που κάνουν αυτή την εκστρατεία για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο την κοινή γνώμη για τα θέματα αυτά που έχουν κεφαλαιόδη χαρακτήρα. και <clears throat> θα ακούσουμε και την κυρία Emma Sankler Webb, η οποία είναι η εκπρόσωπος της Human Rights Watch στην Τουρκία και η οποία έχει εκπονήσει μια έκθεση η οποία βρίσκεται μέσα στην τεκμηρίωσή σας για την σημερινή συνεδρία. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά μαζί με και την παρουσία του πρεσβευτού της Τουρκίας του κυρίου Σαντιμ Γενέλ, τον οποίον ευχαριστώ για την παρουσία του. Του νέου πρεσβευτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στις ε, εργασίες μας εκπροσωπώντας την Τουρκία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον καλωσορίζω. Δουλεύει το διαδίκτυο, η διάδοση στο διαδίκτυο. Πολύ ωραία. <clears throat> Σας προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αχμέτ Ινσέλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα τους λόγους για τους οποίους δεχτήκαμε να είμαστε σήμερα εδώ και τους λόγους για τους οποίους ξεκινήσαμε μια εκστρατεία εδώ και λίγους μήνες για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στην Τουρκία πρώτα, στην Ευρώπη βεβαίως για τα θέματα της καταχρηστικής κράτησης και της ε, ιδιαίτερα διευρυμένης χρήσης της κατηγορίας της τρομοκρατικής δράσης και της συνεργασίας με τρομοκρατικές οργανώσεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Τουρκία για το θέμα του εκδημοκρατισμού και το γνωρίζουμε αυτό. Ανάμεσα στα προβλήματα τίθενται κάποια συγκεκριμένα που συνδέονται με τον εκδημοκρατισμό, κάποια συγκεκριμένα που συνδέονται με την δικαιοσύνη. Αυτά τα δεύτερα είναι, θα έλεγα, στην πρώτη θέση ουσιαστικά σήμερα του ενδιαφέροντός μας. Ιδιαίτερα οι ενέργειες και οι δράσεις που αμφισβητούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνη σε επίπεδο ποινικό. Τρεις νόμοι. Ο ποινικό κώδικας, ο νόμος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η νομολογία, η ποινική νομολογία, είναι θέματα τα οποία έχουν τεθεί επανειλημμένα από την αρχή που ξεκίνησε η Τουρκία να διαπραγματεύεται και να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά της και στα πλαίσια επίσης της προπαρασκευής για το κοινοτικό κεκτημένο. Σε αυτούς τους τρεις νόμους έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, αλλά σήμερα βρισκόμαστε θα έλεγα σε μια κατάσταση η οποία από το 2007-2008 βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι έχει πάει πίσω, ιδιαίτερα στον τομέα της προσωρινής κράτησης, και στον τομέα της κράτησης για τρομοκρατικές ενέργειες ή για την σύσταση εγκληματικών οργανώσεων, συμμοριών σε εισαγωγικά. Τα προβλήματα τίθενται και έχουν υπογραμμιστεί από πολλούς. Καταρχάς μια έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα τις πρώτες μέρες του Γενάρη του Τόμας Χάμερσπεργκ, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών για την Οργάνωση της Δικαιοσύνης και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο υπογραμμίζει τα περισσότερα από τα προβλήματα τα οποία θα σας εκθέσουμε σήμερα πολύ συνοπτικά. Γι' αυτό και η έκθεση του Τόμας Χάμερμπερκ έχει προσαρτηθεί στην παρουσίασή μας και γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσουμε να τη διαβάσετε προσεκτικά γιατί είναι ένας εξαίρετο για τον τρόπο τον οποίο, με τον οποίο η Τουρκία θα ενισχύσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή του νόμου. Πέραν των νόμων βέβαια, Υπάρχει και ένα θέμα νοοτροπίας, ένα θέμα συμπεριφοράς, ένα θέμα ερμηνείας θα έλεγα που θα πρέπει να διέπει τους δικαστές. Κάποιοι νόμοι δεν είναι ακριβώς εύκολα κατανοητοί και δεν μπορούν να εφαρμοστούν με εύκολο τρόπο προς την σωστή κατεύθυνση, προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ποινικέ διαδικασίες, οι οποίες έχουν κάποια σχέση με την πολιτική πλευρά, οι δικαστές αυτόματα θα έλεγα συστρατεύονται με το κράτος εναντίον της κοινωνίας. Και έτσι οι δικαστές διαρμηνεύουν τους νόμους τους συγκεκριμένους προς την κατεύθυνση όχι της κατανόησης των επιχειρημάτων του κατηγορουμένου, όχι του σεβασμού της αρχής της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, αλλά περισσότερο προς την κατεύθυνση της προάσπισης των συμφερόντων που άπτονται με την εθνική ασφάλεια. Ταυτόχρονα οι ποινικέ διαδικασίες στην Τουρκία και ιδιαίτερα οι ποινικέ διαδικασίες οι οποίες εγγράφονται στα πλαίσια του αντιτρομοκρατικού νόμου. Οι ποινικέ αυτές λοιπόν διαδικασίες δεν επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης να υπάρξει μια κατάρτιση φακέλου ανάκριση ισότιμη ανάμεσα στην υπεράσπιση από τη μία και την κατηγορούσα αρχή από την άλλη. Η κατηγορούσα αρχή κατηγορεί και η υπεράσπιση πρέπει να αμυνθεί η κατηγορούσα αρχή δεν λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία και τις αποδείξεις που υπάρχουν και είναι υπέρ του κατηγορουμένου στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυτό καθιστά τις δικαστικές διαδικασίες μακρόσυρτες γιατί η υπεράσπιση δεν μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει παρά μόνο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σε δικαστήριο και όχι κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Το Υπουργείο γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το δικαστήριο γνωρίζει το θέμα της πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών και επανειλημμένα θέλησε να βελτιώσει τις συγκεκριμένες διατεθατίες. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει ανακριτική αστυνομία, η δικαστική μάλλον αστυνομία, και εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει ισότιμα το παιχνίδι ανάμεσα στον εισαγγελέα και την υπεράσπιση από την άλλη ή τον δικαστή και τον δικηγόρο υπεράσπισης, τότε δεν είναι δυνατόν να σμικρινθεί ο χρόνος που διαρκούν αυτές οι διαδικασίες. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα της κράτησης των κατηγορουμένων. Το θέμα της προφυλάκησης, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα, είναι μια πρακτική η οποία θα έλεγα είναι μέσω τιμωρίας αυτόματης εις βάρος των κατηγορουμένων στις περισσότερες δίκες οι οποίες αντιμετωπίζονται στα πλαίσια ε, της εφαρμογής των διατάξεων του αντιτρομοκρατικού νόμου και στα πλαίσια επίσης των διαδικασιών που ακολουθούν τα λεγόμενα ειδικά ποινικά δικαστήρια ή μάλλον ποινικά δικαστήρια ειδικών αρμοδιοτήτων. Οι αλλαγές οι οποίες έχουν ε, υπάρξει στα πλαίσια του αντιμοκρατικού νόμου το 2006 και μετά επιτάχυναν θα έλεγα την χρήση από πλευράς της κατηγορούσας αρχής ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή ακόμα και όταν δεν υπάρχει συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση το να βρίσκεται κανείς σε επικοινωνία με τρομοκρατική οργάνωση και έτσι κατηγορούνται δημοσιογράφοι, κατηγορούνται πανεπιστημιακοί, κατηγορούνται τοπικοί άρχοντες, κατηγορούνται τουρκικής προέλευσης κάτοικοι, κατηγορούνται πολλές φορές αριστεροί ή ακροαριστεροί ή αυτοί οι οποίοι έχουν θέσεις οι οποίες δεν θεωρούνται νόμιμες από την κυβέρνηση ή από ένα τμήμα των αρχών καταστολής, των αρχών ασφαλείας μάλλον. Όλοι αυτοί λοιπόν κατηγορούνται ότι προβαίνουν σε δράσεις στα πλαίσια οργανωμένων συμμοριών ή στα πλαίσια τρομοκρατικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Τουρκία προφυλακίσεις, όχι ε, ιδιαίτερα μακρόχρονες και αυτοί οι προφυλακισμένοι πάρα πολύ συχνά δεν γνωρίζουν για πάρα πολύ καιρό, για μήνες ολόκληρους, ίσως και για ένα χρόνο, καν ποιες είναι οι κατηγορίες για τις οποίες διώκονται και για τις οποίες είναι προφυλακισμένοι. Γιατί, γιατί ο νόμος επιτρέπει στην εισαγγελία να εφαρμόσει την λεγόμενη ειδική διαδικασία απαγόρευσης της πρόσβασης της υπεράσπισης στον φάκελό του. Αν αυτό αφορούσε δύο-τρεις ανθρώπους θα ήταν σοβαρό αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιορισμένα προβλήματα. Όμως όχι. Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι πρακτικές αυτές αυξάνονται συνεχώς εδώ και κάποια χρόνια με πολύ ανησυχητικό τρόπο. Σήμερα, στο τέλος του 10 μάλλον, στην Τουρκία, σύμφωνα με τους αριθμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 8.190 άτομα φυλακισμένοι είναι προφυλακισμένοι ή είναι καταδικασμένοι ήδη, αυτό για ενέργειες που άπτονται της τρομοκρατίας. Ο αριθμός αυτός ήταν 3.335 το 2006 και 3.789-88 το 2004. Τριπλασιάστηκε ο αριθμός αυτός των κρατουμένων λοιπόν τα τελευταία πέντε χρόνια και έχουμε θα έλεγα σε επίπεδο αριθμών έστω, επανέλθει στην θλιβερή κατάσταση την οποία είχε βιώσει η Τουρκία στα πλαίσια της λεγόμενης σκοτεινής περίοδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη δεκαετία του 90, τα τέλη του 90, το 99 σαν παράδειγμα ήταν στη φυλακή τότε άνω των 10.000, 10.330 φυλακισμένοι. Ο αριθμός μειώθηκε πολύ σημαντικά μετά από την αμνηστία του 2000, αλλά σιγά σιγά ξαναφτάσαμε στην ίδια κατάσταση. Και γι' αυτό πλέον κινητοποιούμεθα έτσι ώστε η τουρκική κοινωνία να μην ζήσει για δεύτερη φορά την καταπίεση, την καταστολή, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μπορέσει επιτέλους η τουρκική κοινωνία να είναι μια κοινωνία στα πλαίσια της οποίας οι θεμελιώδεις ελευθερίες γίνονται αντικείμενο σεβασμού Εντοπίσαμε λοιπόν, ακολουθώντας τις εκθέσεις των δικηγορικών συλλόγων, τις εκθέσεις του Τόμας Χάμεσμπεργκ, τις εκθέσεις της, που είναι, ΕΜΑ που είναι δίπλα μου εδώ και επίσης την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επίπεδο προόδου των διαδικασιών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία, εντοπίσαμε λοιπόν κάποια άρθρα του νόμου που άμεσα θα έλεγα βρίσκονται στη βάση αυτών των καταχρηστικών ποινικών διαδικασιών και της υπερβολικής χρήσης και διεύρυνσης ε, της ε, ε, κατηγορίας σύστασης τρομοκρατικής οργάνωσης ή συνεργασίας με τρομοκρατική οργάνωση. Καταρχάς, ο ποινικό κώδικας. Στα πλαίσια του ποινικού κώδικα υπάρχουν δύο άρθρα, το 220 και το 314, το σημείωμα το οποίο σας έχουμε δώσει στη δεύτερη σελίδα έχουμε ε, σε τρεις μικρές παραγράφους υπογραμμισμένα ουσιαστικά τα συγκεκριμένα αυτά άρθρα το 226 με 8 και το 314 του ποινικού κώδικα αφορούν τα συγκεκριμένα αυτά άρθρα το οργανωμένο ή μάλλον το έγκλημα συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση και επίσης μια κατηγορία όταν κάποιος δεν είναι μέλος μπορεί να συνεργάζεται ή να βρίσκεται σε επικοινωνία με τρομοκρατική οργάνωση, κάτι το οποίο περιορίζει και την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία σύστασης ε, πολιτικών οργανώσεων Ο περιορισμός αυτής της ελευθερίας ε, γίνεται χωρίς να υπάρχει συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και θεωρείται η επικοινωνία με τέτοιου είδους οργάνωση έγκλημα ποινικά κολάσιμο. Λοιπόν, το Σύνταγμα συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο άρθρο 6 και 10 περιορίζει την ελεύθερη έκφραση υπεράσπισης. Ο ποινικό κώδικας, κώδικας λοιπόν αυτός, δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα ερμηνεία στον δικαστή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για τις προφυλακίσεις και τις παρατάσεις αποφάσεων που καταδικάζουν σε προφυλακίσεις, αυτά στο άρθρο 10 και στα άρθρα 250 και 252 ο νόμος επιτρέπει την δημιουργία ειδικών έκτακτων διαδικασιών στα πλαίσια των ποινικών δικαστηρίων ειδικού ενδιαφέροντος, ειδικών αρμοδιοτήτων τα δικαστήρια αυτά στην ουσία έχουν αντικαταστήσει τα δικαστήρια ασφαλείας του κράτους που καταργήθηκαν το 2000 μετά από τη σημαντική προσπάθεια που έκανε η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία και μετά από την κινητοποίηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας θυμίζω. Είναι λοιπόν αλήθεια και θα τελειώσω εδώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ευαίσθητο στα προβλήματα τα οποία έχουμε ε, υπογραμμίσει και μάλιστα χθες το απόγευμα η κυβέρνηση παρουσίασε στη Βουλή, στην Εθνοσυνέλευση συγγνώμη, ένα σχέδιο μεταρρύθμισης των συγκεκριμένων άρθρων των νόμων αυτών που έχουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές οι προτινόμενες στον συγκεκριμένο στόχο στοχευμένο θα έλεγα, την βελτίωση της απόδοσης της δικαιοσύνης, της επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών και δεύτερον της διευκόλυνσης της μεταφοράς ποινή για εγκληματικές πράξεις που έχουν σχέση με τον τύπο. Οι αλλαγές αυτές έχουν μεγάλη σημασία για τρεις λόγους σε ό,τι μας αφορά. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα. Το ότι δεν θα φυλακίζεται κάποιος σαν παράδειγμα γιατί έχει ε, εκδώσει ακάλυπτες επιταγές. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν μας αφορά στη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα τα οποία έχουν συγκεκριμένο για μας ενδιαφέρον. Πρώτον, η δυνατότητα μείωσης κατά τα δύο τρίτα των ποινών για πράξεις που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση. Είναι η δυνατότητα που δίδεται στον δικαστή να αξιολογήσει, να εκτιμήσει, ανάλογα με το είδος της αρρωγής προς την τρομοκρατική οργάνωση, να μειώσει την ποινή κατά τα δύο τρίτα. Αυτό αφορά λίγα πρόσωπα, τα οποία επειδή υποτίθεται έγραψαν βιβλία σαν παράδειγμα, μετά από εντολή τρομοκρατικών οργανώσεων βρίσκονται στη φυλακή. Αχμεντ Σίκ σαν παράδειγμα και ο Σενέρ. Αυτοί θα μπορούσαν να απελευθερωθούν χωρίς να θωθούν. Απλά θα μπορούν να βγουν από τη φυλακή γιατί η ποινή τους θα μειωθεί κατά τα δύο τρίτα σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Αλλά μιλάμε εδώ για μία απλή μείωση, μία δυνατότητα μείωση κατά τα δύο τρίτα της ποινής για συγκεκριμένα άμεσα θα έλεγα εγκλήματα, άμεσες ποινικά κολάσιμες πράξεις. Δεύτερον, υπάρχει υποχρέωση να τεκμηριώσουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο οι δικαστές τις αιτιολογικές τους θα έλεγα α, εξηγήσεις σχετικά με τις ποινές τις οποίες επιβάλλουν, ιδιαίτερα σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Σήμερα ο νόμος καθιστά φυσικά τον δικαστή υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να τεκμηριώσει τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις όμως αυτές δεν είναι πολύ συγκεκριμένες και έτσι επιβάλλεται τώρα ο δικαστής να δώσει τρεις συγκεκριμένες απαντήσεις για να τεκμηριώσει έτσι την απόφαση που παίρνει για προφυλάκηση. Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα είναι η κατάργηση της δυνατότητας διακοπής από πλευράς της δικαιοσύνης απαγόρευσης, της απαγόρευσης μιας εφημερίδας, ενός περιοδικού πριν υπάρχει η δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλοφορίας πριν ληφθεί απόφαση από πλευράς του δικαστηρίου. Αυτή επίσης η ρύθμιση είναι σημαντική για μας. Τελειώνοντας, ξαναλέω ότι η μεταρρύθμιση αυτή έχει καλές προθέσεις. Εμπνέεται από καλές προθέσεις. Δυστυχώς όμως οι προθέσεις αυτές δεν έχουν συγκεκριμένες βάσεις. Και μας δίδεται η εντύπωση ότι είναι ένα πολύ διστακτικό βήμα, μισό βήμα, ούτε καν σε σχέση με τη βελτίωση του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. Πιο συγκεκριμένα, για τα θέματα προσωρινής κράτησης και για τα θέματα κατηγοριών που άπτονται τρομοκρατικών ενεργειών. Ο νόμος δεν επιτρέπει να αλλάξει ο ορισμός των συγκεκριμένων ποινικών πράξεων. Είναι πάρα πολύ ευρία η ερμηνεία που δίνεται και τα βήματα τα οποία γίνονται στην ουσία δεν κάνουν πιο συγκεκριμένη τη διαδικασία, Πρόκειται για μία θα έλεγα καλοπιστική αν θέλετε βελτίωση και όχι βελτίωση επί της ουσίας. Η Τουρκία βέβαια είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και γι' αυτό ζητάμε οι υποχρεώσεις της Τουρκίας. Οι εδραζόμενες στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης να γίνονται αντικείμενο πλήρου σεβασμού. Η μεταρρύθμιση αυτή μόνο εν μέρη και με περιορισμένο τρόπο ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις ε, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης στην Τουρκία. Συνεπώς ζητάμε οι Ευρωπαίοι φίλοι να πάρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέρος στην προσπάθεια βελτίωσης της σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Έχει κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία μια κοινωνία των πολιτών η οποία ανησυχεί πάντα για καταχρηστική χρήση από πλευράς της δικαιοσύνης πρακτικών προφυλάκησης απαράδεκτων και δεν θέλουμε η Τουρκία να γίνει κάτι το οποίο είχαμε γνωρίσει τα μολυβένια χρόνια, όπως λέγαμε κάποτε, όπως έλεγαν και οι Ιταλοί τη δεκαετία του 80. Ευχαριστούμε πολύ Ινσέλ, νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά τα έχετε θέσει με μεγάλη σαφήνεια, κάτι το οποίο θα επιτρέψει μια συζήτηση τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ακίνα Ταλάη. Είπα προηγουμένως ότι είσαστε μια σημαντική προσωπικότητα της ε, Ένωσης των Δικηγόρων για το Ποινικό Δίκαιο. Είσαστε δικηγόρος και είσαστε ο δημοσιογράφος των δύο δημοσιο... είσαστε ο δικηγόρος συγγνώμη, των δύο δημοσιογράφων που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία μας ad hoc το Νοέμβριο για τον κύριο Αχμέτ Σιτ και τον Εντίμ Σενέρ. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διόρθωση πρώτα. Δεν είμαι δικηγόρος του Νεντίμ Σενέρ αλλά του Αχμέτ Σίκ μόνο. Έχω όμως πολλούς άλλους πελάτες εντολής, ε, επίσης δημοσιογράφους και μάλιστα ένας από αυτούς είναι πολύ γνωστός και μάλιστα συναδελφός σας ως ε, βουλευτής, ο Μουσταφά Μπαλμπάη και άλλος στο ΣΕΛΕΚ. Άρα ε, εκτελώ χρέη συνηγόρου και αυτών των κρατουμένων δημοσιογράφων και βουλευτών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των δύο χωριστών δικών των πελατών μου, των εντολέων μου, είδα πολλά πράγματα τα οποία έχω έρθει να σας παρουσιάσω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο παραδείγματα, τους δύο δημοσιογράφους, τον οποίον ο πρώτος εξελέγει στι προηγούμενε εκλογέ, τι τελευταίε εκλογέ, με το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται για τον δημοσιογράφο στο Φαμπαρμπάι, Ενώ ο άλλο είναι ε, ο κρατούμενο, ε, επειδή έγραψε ένα βιβλίο, ο Αχμέτσικ και όπως είπα βρίσκεται ακόμη ε, στη φυλακή κρατούμενος, προφυλακισμένος. Ανέλαβα λοιπόν ε, να τους υπερασπιστώ, την υπερασπισή τους από τη στιγμή που προσήχθησαν ε, στην αστυνομία και είμαι ε, από πρώτο χέρι μάρτυρα των όσων έχουν περάσει. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν είμαι σε θέση να εκτελέσω το έργο μου ως συνήγορος υπό τις συνθήκες που επικρατούν, η απάντηση που θα σας δώσω είναι ρητά όχι. Διότι και οι δύο αυτοί δημοσιογράφοι δικάζονται όχι με τακτικούς κανόνες, με το τακτικό δίκαιο δηλαδή της εξαγωγής της δίκης, αλλά με έκτακτους κανόνες, με ειδικού κανόνες. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία και κατά την ανάκριση δεν μπόρεσε να ασκηθεί η λειτουργία του συνηγόρου. Μόνο παθητικά ήμουν παρόν, ως μάρτυρας, ούτως υπήν, στη διαδικασία αυτή, που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Και όταν μετά από πολλούς μήνες άρχισε η δίκη, με πολύ περιορισμένο τρόπο μπόρεσα να ασκήσω το λειτουργήμά μου ως συνήγορος. Να σας πω λοιπόν πώς διεξάγεται αυτή η δικασία. Εν γέννη, τις πρώτες πρωινές ώρες, νωρίς νωρίς, γίνεται επιδρομή στο σπίτι του υπόπτου από την αστυνομία. Γίνεται έρευνα κατοίκων συλλέγονται τα βιβλία τους, οι σημειώσεις τους, χιλιάδες σελίδες, οι ηλεκτρονικοί τους υπολογιστές κατάσχονται. Ο συνήγορος ρωτάει ποιος είναι, ποια είναι η κατηγορία, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Η απάντηση είναι τρεις-τέσσερις λέξεις μόνο. Ότι ε, κατηγορείται για συμμετοχή στην, σε τρομοκρατική οργάνωση. Δεν δίνεται δηλαδή καμιά άλλη απάντηση πέραν αυτών των ολίγων λέξεων. Στη συνέχεια. Ρωτάμε τι αποδείξεις έχετε γι' αυτό. Πάλι συνοπτική απάντηση ότι έχει ληφθεί απόφαση για περιορισμένη πρόσβαση και για απαγόρευση πρόσβαση στο σχετικό φάκελο και ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς ούτε να δει αποδεικτικά στοιχεία, ούτε να τα διαβάσει, ούτε να πάρει αντίγραφο. Εν γέννη δε, η πρακτική είναι ότι μένει ο κατηγορούμενο για τέσσερι μέρε στο κρατητήριο, ε, στο αστυνομικό τμήμα δηλαδή. Μέσα αυτέ τι τέσσερι μέρε τι συμβαίνει. Οτιδήποτε έχει ε, συλλέξει αστυνομία από το σπίτι του υπόπτου, ε, έγραφα σημειώσεις, ε, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αναλύονται και χρησιμοποιούνται για την διατύπωση της κατηγορίας. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται η σύλληψη και η προσαγωγή, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Απλώς είναι πολύ σίγουρη η αστυνομία ότι με την σύλληψη θα βρει ταυτόχρονα και στο σπίτι του ε, υπόπτου, του δημοσιογράφου, πάρα πολλά στοιχεία και αρκετά για να τον κατηγορήσει στη συνέχεια. Γίνεται η ανάκριση, η απολογία και εν γέννη χωρίς ίσως μόνο κάποιες εξαιρέσεις να υπάρχουν, προσάγεται ενώπιον του δικαστού, ο οποίος ε, ρωτάει μόνο την εξή ερώτηση στον ύποπτο, τον κατηγορούμενο. Κατηγορήστε για συμμετοχή σε τρομοκρατική ε, οργάνωση, απολογηθείτε. Αυτό του λέει μόνο. Τι μπορεί λοιπόν να πει κανείς σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να ρωτήσει πού είναι οι αποδείξεις πάνω σε οποίες στηρίζεται αυτή η κατηγορία. Πείτε μου ποιε είναι να μπορέσω να τις απαντήσω, να τις αντικρούσω, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όχι. Η απάντηση έρχεται και πάλι ότι είναι απόρριτα τα στοιχεία, απόρριτα τα αποδεικτικά και μέχρι να ξεκινήσει η ε, δίκη ε, δεν υπάρχουν δεν υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί κανείς για, ε, για τα στοιχεία του φακέλου. Στη συνέχεια και πολύ αφηρημένα, με πολύ αφηρημένους όρους, ε, γιδίδεται η απόφαση για την προσωρινή κράτηση, στην οποία και πάλι με πολύ αφηρημένους όρους, με όρους ε, επαναλαμβανόμενους, απορρίπτεται οποιαδήποτε αίτηση για αποφυλάκηση. Στην περίπτωση του Μουσταφά Μπαλμπάη για να ολοκληρώσω την υπόθεση αυτή, θέλω να σας πω ότι είναι ακόμη προφυλακισμένος. Τρία χρόνια έχουν περάσει. Είναι στο τέταρτο χρόνο της προφυλάκησής του. Και νομίζω ότι στην ιστορία του, της ανθρωπότητας ολόκληρης δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Κάθε μέρα ξεκινάει μια δίκη από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνεχίζεται την άλλη μέρα. Έχουν γίνει ήδη 150 δικάσιμοι. Είμαστε στην 152η σήμερα που βρίσκομαι εγώ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Και μέχρι στιγμής, με όσε ώρες και να κρατήσει αυτή η δικάσιμος, κάθε φορά ξαναγυρνάμε από την αρχή. Από την ε, αρχή δηλαδή της, ε, των ερωτήσεων της ανάκρισης. Αυτό για να σας εξηγήσω πόσο, με πόσους βραδείς ρυθμούς προχωράει αυτή η δίκη. Και πάλι ως προς την προσωρινή κράτηση, λόγος κράτησης δεν δίνεται, δηλαδή προβάλλεται η αιτιολογία ότι δεν έχουν ακόμη συλλεχθεί υπαρκή στοιχεία αποδεικτικά και ω εκ τούτου πρέπει να παραμείνει προφλεξιτέως ο κατηγορούμενος. Ο άλλο μου πελάτη, ο Σουκ, ε, συνελήφθη το Μάρτιο που μας πέρασε και πάλι πέρασε από την ίδια διαδικασία. Μετά την ε, κράτηση, αφού μάλλον συνελήφθη, πέρασαν 24 ώρες για να δει το, δικηγόρο του, έμεινε στο κρατητήριο της φυλακής, μετά προσήχθη στον ε, ε, ανακριτή την προσωρινή του κράτηση και, και πάλι δεν μπόρεσε να ενημερωθεί για τους λόγους για τους οποίους ε, κατηγορείται και θεωρείται προφυλαξιστέως. Μετά λοιπόν την προφυλάξη, την ε, απόφαση για την προσωρινή κράτηση, έγιναν ε, πολλές εκδηλώσεις και έντονες αντιδράσεις εκφράστηκαν γενικότερα από την κοινή γνώμη ένας αρκετά γνωστός ε, για το ανακριτικό του έργο εισαγγελέα ε, δημοσίευσε το εξής κείμενο όπου λέει ότι ο Αχμέτσικ δεν κατηγορείται για το βιβλίο αυτό το οποίο είχε ετοιμάσει αλλά για ε, εγκλήματα των οποίων τα αποδεικτικά παραμένουν απόρριτα και κρυφά για να διεξαχθεί ομαλά η δίκη και για λόγους εξαγωγής της δίκης. ότι έχει προσπαθήσει να επηρεάσει την έκβαση της δίκης του, ότι αυτό το ίδιο πράγμα είναι, αποτελεί και έγκλημα, ότι έχει προσπαθήσει να εξυπηρετήσει σκοπούς τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι... και ότι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι αυτή η υπόθεση είναι πάρα πολύ ε, λεπτή και να, όλοι οι δημοσιογράφοι να την παρακολουθούν με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή, τόσο ο Αχμέτσικ όσο και ο Νεντίμ Σενέρ που συνελήφθη ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να απασχολούν τους δημοσιογράφους. Αυτό το μήνυμα δηλαδή του ανακριτή Παύλα Ισαγγελέα ε, ουσιαστικά λεγόταν στους υπόλοιπους δημοσιογράφους προσέξτε μην ασχοληθείτε με το θέμα αυτό διότι κινδυνεύετε να πάθετε τα ίδια. Και όχι μόνο αυτό. Ελήφθη ταυτόχρονα απόφαση να απαγορευτεί η δημοσίευση του βιβλίου και να κατασχεθούν όλα του τα αντίγραφα ή αντίτυπα από την αστυνομία. Έτσι λοιπόν έλαβε απόφαση ο ανακριτής Παύλα εισαγγελέα ότι ακόμη και το ένα μοναδικό αντίγραφο που είχαν στα χέρια τους οι συνήγοροι του Αχμέτσικ θα έπρεπε να παραδοθεί, διότι ήταν αντικείμενο ή αποδεικτικό εγκληματική ενέργεια. Και άρα θα έπρεπε να το παραδώσουν οι συνήγοροι στην αστυνομία. Εάν δεν αρνούνταν να το πράξουν, θα κατηγορούνταν για σύμπραξη με τρομοκρατική οργάνωση και θα προσάγονταν στη δικαιοσύνη. Αυτά όλα με επίσημα έγραφα. Ταυτόχρονα πολλοί από τους ε, δικηγόρους που είχαν αναλάβει καθήκοντα στην υπόθεση του TV, του, της ιστοσελίδας ε, της δημοσιογραφής, ΚΙΣ, βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση με αποφάσεις για ε, κατάσχεση των αντιτύπων που, που παρά τις αντιδράσεις τους τελικά αναγκάστηκαν να παραδώσουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των βασικών όρων άσκησης του λειτουργήματός μας. Την ίδια μέρα απέστειλα αίτησα, αίτηση στο, ε, στην Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Τουρκίας ζητώντας να με στηρίξουν διότι αυτή η απόφαση που είχε ληφθεί η κατάσχεση ακόμη και των βιβλίων αποτελούσε σημαντική παραβίαση των ε, δικαιωμάτων της, ε, των συνηγόρων της υπεράσπισης. Αυτό το θέμα βέβαια πήρε διαστάσεις και στην Τουρκία ολόκληρα και στη διεθνή κοινότητα. Και κατόπιν αυτού ε, τέθη τέρμα έπαυσε στα ξαφνικά η απόφαση αυτή, η προσπάθεια για κατάσχεση όλων αντιπτύπων. Και προχωράμε στον Αύγουστο, όπου ξεκίνησε η δίκη, όπου και πάλι αντιμετώπισα ένα παράδοξο. Κοιτώντας το φάκελο, διαπιστώνω, το φάκελο της υπόθεσης, διαπιστώνω ότι ε, υπάρχει κατηγορία εις βάρος του Αχμέτσικ, υπάρχουν κατηγορίες στηριζόμενες σε υποκλοπή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Αχμετσίκ με τους δικηγόρους του, με τους συνηγορούς του. Ο κατηγορούμενος λοιπόν δεν μπορεί να έχει απόρριτη συνομιλία με τον δικηγόρο του. Αυτό αποτελεί βασική αρχή, όχι μόνο οικουμενική του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας, αλλά και στη χώρα μας κανονικά. Έχει, ε, έχει θέση, έχει εγγραφεί στην νομοθεσία μας. Ζήτησα λοιπόν αμέσως ε, να αφαιρεθούν αυτά τα στοιχεία των, ε, οι απομαγνητοφωνίες των τηλεφωνικών διαλέξεων από τον ε, φάκελο της κατηγορίας, του κατηγορητηρίου και να καταστραφούν, διότι ταυτόχρονα αποτελούν και εμπόδιο στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και σε τελευταία ανάλυση κάποιου τύπου απειλή. Το ζήτησα αυτό πριν από μερικές μέρες, λίγο πριν έρθω εδώ δηλαδή, αλλά απερίφθη αυτή η αίτηση. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η ανάκριση στην υπόθεση του Αχμέτσουκ. Εμείς ε, συνεχίζουμε τα καθήκοντά μας να τα ασκούμε ως ε, ε, συνήγοροι. Και αυτό που παρατηρώ, για να ολοκληρώσω, είναι ότι ιδιαίτερα την υπόθεση της τρομοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία δεν είναι καθόλου σαφή τα όρια τι είναι τρομοκρατία και την ελευθερία έκφρασης οι δε ε, εισαγγελείς και δικαστές δεν συμπεριφέρονται με την ευαισθησία και την προσοχή που απαιτείται στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Τουναντίον ε, συγχέουν τα όρια και διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της ε, κατηγορίας τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νομίζω ότι η συγκεκριμένη αυτή η πρακτική που αναφέρατε ως δικηγόρος ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική για μας. Η τελευταία παρέμβαση, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη, ο οποίος ίσως θα θέλει και αυτός να αναφέρει τι ακριβώς ε, διακυβεύεται στην δικαστική μεταρρύθμιση και είναι ακριβώς και η πρώτη ευκαιρία που έχει σήμερα για αυτή την πρόταση η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα θα μας εξηγήσετε ενδεχομένω με ποιο τρόπο μπορεί να άρει ορισμένα από τα προσκόμματα στην ελευθερία έκφραση τα οποία αναφέρθηκαν. Θα ήθελα να δώσω λόγο στην κυρία Έμα Έμα Βέμπ για από την Human Rights Watch και η οποία είναι η συντάκτρια μιας έκθεσης που έχετε όλοι στο φακελό σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που οι συνάδελφοί μου σταμάτησαν. και να αφηγηθώ λίγα και την ιστορία των περασμένων χρόνων για το πώς ο αριθμός των ποινικών διώξεων βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου στην Τουρκία αυξήθηκε σημαντικά και πώς αυξήθηκε και ο αριθμός των ατόμων τα οποία ε, προφυλακίστηκαν και τριπλασιάστηκε ουσιαστικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η ύποπτοι αδικημάτων τρομοκρατίας που βρίσκονται σε προφυλάκηση το 2008 βρισκόταν γύρω στις 3.000, ενώ τώρα είναι τριπλάσιος αυτός ο αριθμός, έχει φτάσει τα, 9.000 προφυλακισμένων. Είναι πολύ σημαντική αύξηση και θα ήθελα να περιγράψω τους νόμους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και τα σχήματα διώξεως που είδαμε να ασκούνται τα προηγούμενα χρόνια αυτή η πρακτική βασίζεται σε πολλά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν στην Τουρκία για την έλλειψη δίκαιας διοικής που έχουν αναφερθεί και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε επανειλημμένες αποφάσεις. Είναι το θέμα του, της διάρκειας της ε, δικαστικής διαδικασίας που είναι μόνιμο πρόβλημα στην Τουρκία και επίσης του θέματος της αυθαίρετης προφυλάξης, αυθαίρετης κράτησης και προφυλάξης. Αυτά είναι τα άρθρα 6 και τρία, όπου υπήρξαν προβλήματα στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν από το παρελθόν, δεν είναι προβλήματα που παρουσιάστηκαν μόνο πρόσφατα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η χρήση της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, η ευρεία χρήση της νομοθεσίας για την τρομοκρατία φαίνεται πολλές φορές στην, από έξω ότι στρέφεται μόνο κατά των δημοσιογράφων και ότι μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να πω όμως ότι δυστυχώς είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα αυτό. Δεν είναι μονάχα οι δημοσιογράφοι, αλλά είναι και πολύ ευρύτερε ομάδε του πληθυσμού που θίγονται από αυτή την νομοθεσία. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα στην Τουρκία που κράτησε δύο χρόνια, προσπαθώντα να δούμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται η νομοθεσία περί τρομοκρατίας κατά των ατόμων που διαμαρτύρονται σε μια διαδήλωση, παραδείγματο χάρη. Είναι άτομα τα οποία συμμετέχουν σε διαδηλώσει οι οποίε μπορεί να γίνουν βίε. Κάποιοι πετάνε πέτρε, μερικέ φορέ πετάνε και κοκτέιλ μολότοφ. Και επίση πολλέ φορέ φωνάζουν συνθήματα που θεωρούνται επιλήψιμα. Η διαχείριση αυτών των διαδηλώσεων σε καμιά κοινωνία δεν είναι εύκολη. Αλλά η νομοθεσία η οποία άρχισε να σε αυτούς τους ε, διαδηλωτές, η πλειοψηφία των οποίων ήταν Κούρδοι, ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληροί νόμοι αντιτρομοκρατικοί, γιατί κατηγορήθηκαν και διώχθησαν σαν να ήταν μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο νόμοι, το, η διάπραξη αδικήματος για λογαριασμό τρομοκρατικής ε, ε, οργάνωσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο επισύρει την ίδια ποινή όπως το να είναι κανείς μέλος μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι βαριές οι ποινές που επισύρονται, 7,5 χρόνια με πρόσθετες ποινές οι οποίες μπορούν να προσθεθούν για, βί, για βίαιες ενέργειες. Το να είναι κανείς μέλος λοιπόν σε μια τρομοκρατική οργάνωση να εξισωθεί με ένα μέλος τρομοκρατικής ε, ε οργάνωσης, σε αυτό προστίθεται η χρήση βίας. πραγματικά χάρη το να πετάξει κανείς πέτρες και επίσης τα συνθήματα που φωνάζει κανείς ως χρήση προπαγάνδας. Μπορεί να φτάσει κανείς σε αστρονομικούς αριθμούς σε συνολική ποινή λόγω αυτών των θεμάτων. Εμείς έχουμε τονίσει ότι δεν υποστηρίζουμε την χρήση βία στις ε, διαδηλώσεις και δεν συγχωρούμε τη χρήση βίας σε διαδηλώσεις. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν νόμοι κατά των ε, βίαιων ενεργειών σε διαδηλώσεις, για την καταστροφή περιουσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής, όλα αυτά περιουσία, το οποίο μας ενδιέφερε περισσότερο ήταν περιπτώσεις όπου η μόνη παρουσία και μόνο σε μία διαδήλωση και όχι βίαιες ενέργειες <clears throat> μπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου με μεγάλες περιπτωσει οπου Πριν από δύο χρόνια υπήρξε μια μεγάλη εκστρατεία στην Τουρκία για τα θέματα αυτά γιατί ανήλικοι μπορούσαν και αυτοί να υφίστανται τέτοιου είδους διώξεις. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός που να μην επιτρέπει τη χρήση αυτής της νομοθεσίας για ανηλίκους. Αυτό καταργήθηκε. Αλλά δεν έχει λυθεί η ουσία του προβλήματος που είναι το γεγονός ότι η διαμαρτυρία μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατική ενέργεια. Για μας αυτό είναι ένα πάρα πολύ προβληματικό θέμα, το οποίο ισοδυναμεί με ένα περιορισμό στο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είδαμε μια μεγάλη αύξηση της χρήσης αυτών των νόμων, όχι μονάχα εναντίον διαμαρτυρώμενων σε διαδηλώσεις, αλλά γενικά κατά ακτιβιστών, κυρίως Κούρδων ακτιβιστών, αλλά εναντίον και άλλων πολιτικών ακτιβιστών, ε, φοιτητών, δημοσιογράφων. Ευραία λοιπόν στρώματα του πληθυσμού έχουν πληγεί από αυτή, της, από αυτή την νομοθεσία. Κυρίως όμως είναι Κούρδοι ακτιβιστές οι οποίοι θεωρούνται ότι πρόσκυνται ιδεολογικά με το ΠΚΚ, το, την οργάνωση αυτή η οποία θεωρείται τρομοκρατική. Η, η αυξημένη λοιπόν προσφυγή σε αυτούς τους νόμους τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει και σε μια συνολική καταστολή στους Κούρδους πολιτικούς κουρδικούς ακτιβιστές εναντίον, εναντίον των Κούρδων πολιτικών ακτιβιστών με την κατηγορία ότι ανήκουν σε μια υποτιθέμενη πολιτική πτέρυγα του ΠΚΚ, τη λεγόμενη KCK, την Ενότητα Κουρδικών Κοινοτήτων και υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει μια σύνδεση αυτών οι οποίοι συμμετέχουν σε αντίστοιχους πολιτικού κύκλου μεταξύ μεταξύ των οργανώσεων αυτών μεταξύ τους και, μεταξύ, και με την τρομοκρατική αυτή οργάνωση, το ΠΚΚ. Αυτό οδήγησε σε ενέργειες καταστολής που οδήγησαν στη σύλληψη εκατοντάδων και χιλιάδων ακόμα ατόμων τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των ομάδων οι οποίες έχουν ε, τύχη δίωξη είναι πολλές φορές και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είδε πολλούς από τους ηγέτες των τοπικών του της παρατημάτων στο νοτιοανατολική Τουρκία και κάποια άτομα από το διοικητικό του συμβούλιο να ε, φυλακίζονται. Ο Μουχάμετ Έρμπεϊ, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος του Διάρμπακερ, έχει, είναι ήδη δύο χρόνια στη φυλακή. Ο, επικεφαλής λοιπόν της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ανατολική Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μονάχα το θέμα της παρατεταμένης προφυλάξης και αυθαίρετης πολλέ φορέ προφυλάξη, αλλά και η χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου και η αυθαιρεσία στην ε, ε, απαγγελία κατηγοριών είναι στοιχεία τα οποία βάσει του, μέσα στο, στη διεθνή Τάξη θα ήταν πάρα πολύ αδύναμα αποδεικτικά στοιχεία, πάρα πολύ ασαφή και αδύναμα στοιχεία για να κατεδικαστεί κάτω. Αν δούμε λοιπόν την τουρκική νομοθεσία, τον ποινικό κώδικα και τον αντιτρομοκρατικό νόμο, θα πρέπει να δούμε καλύτερα ποιο είναι ο ορισμό τη τρομοκρατία και να εξασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί με αυτόν τον ευρύτατο τρόπο σε άτομα τα οποία δεν έχουν διαπράξει πράξεις οι οποίες σύμφωνα με, την, με το διεθνές δίκαιο είναι τρομοκρατικές ενέργειες, δηλαδή ενέργειες που οδηγούν σε θανάτωση ατόμων σε απαγωγές ομήρων, σε άμεση προτροπή προς ε, χρήση βίας ή φυσικά σε παροχή υλικής υποστήριξης για μια παράνομη ενόπλη τρομοκρατική οργάνωση. Όλα αυτά είναι δραστηριότητε οι οποίε θεωρούνται τρομοκρατικέ ενέργειε στι χώρε μα. Αλλά αυτή τη στιγμή στο τουρκικό νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει τέτοιου είδου περιορισμό στο τι αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια και η γενικότητα στις κατηγορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να καταπολεμήσει κανείς την τρομοκρατία. Όταν εφαρμόζει τον αντιτρομοκρατικό νόμο σε μια όλο και διευρυνόμενη ομάδα του πληθυσμού, αυτό δεν αντιμετωπίζει τις θεμητές ανησυχίες που μπορούν να υπάρχουν για την ύπαρξη τρομοκρατίας. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν δώσει σε σχέση με την εφαρμογή τη δικαιοσύνη στην Τουρκία. Το να φωνάσει κανεί κάποια συνθήματα, αυτό μπορεί να ακόμα και αυτό αν είναι ε, βίο, το σύνθημα δεν σημαίνει ότι είναι προτρόπη σε βία. Στην περίπτωση Γκιούλε αντίον τη Τουρκία πριν από 2-3 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΕΔΑ, το ανέφερε αυτό, ότι αυτό πρέπει να περιληφθεί στην ελεύθερη έκφραση απόψεων. Υπάρχουν λοιπόν οι κατευθυντήριε γραμμέ του ΕΔΑΔ και οι ελπίδε μα είναι ότι θα υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειε από την τουρκική κυβέρνηση και θα μπορέσει να εισαγάγει διατάξει στην νομοθεσία που λένε ότι βία ενέργεια είναι μια ενέργεια η οποία είναι, αποτελεί προτροπή στη χρήση βία και αλλιώ δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπινη πράξη. Αυτό προ το παρόν δεν υπάρχει στην τουρκική νομοθεσία. Στρέφομαι τώρα στα πάρα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία σχεδιάζει να εφαρμόσει η τουρκική κυβέρνηση. Είναι ένα μεγάλο πακέτο ε, δικαστικής μεταρρύθμισης. Δεν έχουμε εξετάσει όλα τα στοιχεία αυτού του πακέτου που θα περάσει και από την Νομική Επιτροπή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Κατα... Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα τα οποία πρέπει να τα χαιρετήσουμε και να τα καλωσορίσουμε μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπήρξε η απόφαση ότι δεν μπορούν να ε, κατάσχονται και να αναστέλλεται η κυκλοφορία περιοδικών γιατί αυτό ισοδυναμεί με λογοκρισία για λόγους καταπολέμησης τρομοκρατίας. Φαίνεται ότι αυτό λοιπόν θα καταργηθεί και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Υπάρχει επίσης το θέμα της αναστολής των ε, διώξεων και των ανακρίσεων έναντι αυτών που είναι υπόδικοι, μάλλον είναι υποκατηγορία για, για αδικήματα που επισύρουν ποινές κάτω από πέντε έτη. Αυτό θα ελαφρώσει το ποινικό σύστημα, θα απελευθερωθούν κάποιοι κρατούμενοι, κάποιες ε, ποινές θα ανασταλεί η έκτησή τους. Όλα αυτά μπορούν να είναι πολύ θετικά και σημαντικά βήματα. Αλλά υπάρχει και ένα εάν Υπάρχει μη προϋπόθεση ότι δεν πρέπει κανείς να, να, ε, να επαναλάβει το ίδιο αδίκημα μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό όμως είναι και ένας τρόπος να καταστήλει κανείς την ελευθερία έκφρασης με το πρόσχημα της υποτροπής. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα της μη αυτόματης παράταση τη προφυλάξη τη προσωρινή κράτηση. Αυτή τη στιγμή τα δικαστήρια το πράττουν αυτό χωρί να εξετάσουν πραγματικά το φάκελο, χωρί να δώσουν στου ε, κρατούμενου κάποια δυνατότητα ουσιαστική προσφυγή. Αν υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, θα είναι καλύτερα, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και αυτό θα είναι ένα μήνυμα προ τα δικαστήρια να είναι πιο προσεκτικά στην επιχειρηματολογία με την οποία παρατείνουν την προφυλάξη. Κατανοούμε όμω ακόμα ότι υπάρχουν κάποια αδικήματα, τα λεγόμενα εγκλήματα καταλόγου, είναι πολύ δύσκολο να το αναφέρει αυτός, αλλά υπάρχει ένας κατάλογος θετικός αδικημάτων για τα οποία η απόφαση για την παράταση της προφυλάκησης είναι σχεδόν αυτόματη και αυτό φυσικά περιλαμβάνει τα εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν στο νόμο περί της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να πω επίση ότι είναι σημαντικό για την τουρκική κυβέρνηση να λάβει υπόψη <clears throat> τι ιδιαίτερα σαφεί προτάσει που περιέχονται στην έκθεση του Τόμα Χάμαρμπεργκ για την ε, εφαρμογή της δικαιοσύνης και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αυτό είναι μια θαυμάσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές για, το, για τα σημεία που πρέπει να υπάρξει βελτίωση στο νομικό και δικαστικό σύστημα της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει δημιουργήσει ένα ειδικό χάρτη για τη δικαστική μεταρρύθμιση στην πρόσφατη έκθεση πρόοδου της από το τέλος του 2011 είναι η ελπίδα μας ότι η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα αυτό και να εξασφαλίσει ότι μέσα στο νομικό σύστημα τρομοκρατική ενέργεια είναι μια βία ενέργεια, μια προτροπή σε βία ή μια υλική υποστήριξη προς μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό πρέπει να φαίνεται σε έμπρακτες ενέργειες και όχι μονάχα σε έκφραση άποψης ή στην χρήση του νόμιμου δικαιώματος του συνέχεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν αιτία δίωξη για, το, για τρομοκρατία. Ευχαριστώ κυρία Σέγκρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα. Κάποιος θέλει το λόγο μπορεί να τον ζητήσει. Αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πρέσβη για να αναφερθεί και αυτό σε αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων το οποίο παρουσιάστηκε χθε και σήμερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Ήταν μαζί μας την τελευταία συνάντηση ο Υπουργός Δικαιοσύνη. Θα προσκληθεί επίση και στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης και σίγουρα θα επανέλθει σε αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν σημαντικά βήματα πάνω σε θέματα τα οποία έχετε ήδη θέσει αλλά μιας και κατετέθησαν σήμερα οι προτάσεις αυτές, είναι προφανές ότι η δική σας παρέμβαση ίσως μπορέσει να μας φωτίσει λίγο για να δούμε αν πράγματι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο σήμερα ανάμεσά σας. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μου και είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος του τύπου της τηλεόρασης, των μέσων ενημέρωσης, είναι μια βασική μας ανησυχία. Αν πράγματι εμείς πούμε σαν Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε, ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα, θα το αντιμετωπίσουμε για να ανακάμψει η κατάσταση. Μιλάμε για την μεγάλη διάρκεια των δικών, μιλάμε για προβλήματα που υπάρχουν στην απονομή δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να επανεξεταστούν. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ομάδα παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων. Γιατί? Γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία βαθιάς μεταρρύθμισης της χώρας και πολιτικής μεταρρύθμισης και οικονομικής μεταρρύθμισης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτικές μεταρρυθμίσεις αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η ομάδα αυτή συναντάται πάρα πολύ συχνά και στην τελευταία συνάντηση στην οποία πήρα μέρος στην Κόνια το Δεκέμβριο, στο Εικόνιο συγγνώμη το Δεκέμβριο, τα θέματα αυτά συζητήθηκαν σε βάθος. Αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι κάποιες πρώτες ιδέες και είναι σαφές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε την αρχική του πρόταση στις 19 Ιανουαρίου, το κατέθεσε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και το γραφείο του Πρωθυπουργού χτες το επέστρεψε στο Κοινοβούλιο. Αυτό δείχνει τελικά την ταχύτητα και την αίσθηση του κατεπήγοντος που έχει το θέμα αυτό. Θα πρέπει να το, αποφασί... να το αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τι προβλέπει τώρα η ρύθμιση αυτή. Αυτά τέθηκαν και από τον καθηγητή κ. Ίνσελ. Νομίζω ότι βασικά αυτό το σχέδιο νόμου καλύπτει τις περισσότερες από τις ανησυχίες ακούστηκαν εδώ. Θα τροπολογήσει πολλούς νόμους του ποινικού κώδικα, της ποινική διαδικασίας, της νομολογίας. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να πω ότι οι προθέσεις του νόμου αυτού είναι σωστές δεν είναι ένα διστακτικό βήμα. Θέλουμε να απομακρύνουμε τις δυσκολίες αυτές, ακούμε τις δυσκολίες αυτές όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ε, τουρκικό. Οφείλουμε να λύσουμε το θέμα αυτό από μόνοι μας. Η ομάδα, μεταρρύθμισης των, η ομάδα μάλλον παρακολούθησης των ε, εποπτείας των μεταρρυθμίσεων θα συναντηθεί ξανά τον Μάρτιο. Ε, όπως σας είπα, εστάλει από το γραφείο του Πρωθυπουργού στην Εθνοσυνέλευση η πρόταση. Απαιτείται κάποιος χρόνος. Μέσα σε δύο μήνες ελπίζω να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό επιθυμούμε και αυτό ελπίζουμε να γίνει. Όταν εφαρμοστεί ο νόμος αυτός πλήρως, τότε θα, θα αφορά δύο εκατομμύρια περιπτώσεις. Κάποιες είναι απλά παραπτώματα, αλλά κάποιες άλλες είναι σημαντικότατα θέματα. Η πρόταση νόμου δεν είναι τέλεια, προφανώς, αλλά η πρόθεση και η τάση είναι σωστή. Να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και μία δεκαετία στην Τουρκία υπήρχε η θανατική καταδίκη και έχουμε φύγει από εκεί. Ακολουθούμε λοιπόν μία θετική πορεία. Δεν έχουμε ξεπεράσει τις δυσκολίες, γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτήν την Επιτροπή Εποπτείας των Μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Το ένα είναι η νομοθεσία και το άλλο η εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε επίπεδο νομοθετικό οι διαδικασίες συνεχίζονται. Και όταν λέμε συνεχίζονται, ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα τα οποία είναι πηγή ανησυχίας του λαού μας, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτή την περίπτωση είναι η εφαρμογή του νόμου. Και γι' αυτό ακριβώ και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπαιδεύουμε, καταρτίζουμε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους για το πώς πρέπει να ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση γιατί έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο, όπως ακούσαμε, αντιμετωπίζουν την διαδικασία οι δικαστές. Αν η νομοθεσία είναι τέλεια και η εφαρμογή ατελής, το πρόβλημα παραμένει. Και γι' αυτό ακριβώς ε, συναντάται τακτικά και εξετάζει προσεκτικά τα θέματα η Επιτροπή Εποπτείας των Μεταρρυθμίσεων. Σας είπα ότι οι τάσεις ε, που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην τουρκική κυβέρνηση είναι θετικές Κάποιοι είπατε ότι είναι ημίμετρα. Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι πλήρη τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε και θέλουμε να καλύψουμε όλων τις ανάγκες. Τελειώνοντας να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δυστυχώς τρομοκρατία υπάρχει και η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να φροντίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φροντίζοντας όμως και την ασφάλεια των πολιτών. Κάθε κυβέρνηση στον κόσμο αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτό πρέπει να κάνει και η τουρκική κυβέρνηση και αυτό θα κάνει. Νομίζω ότι ακολουθούμε ένα σωστό δρόμο. Βέβαια δεν έχουμε ξεπεράσει όπως είπα τις δυσκολίες, δεν έχουμε φτάσει στην τελική φάση, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όταν τελειώσει η διαδικασία όλοι θα είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά για τις διευκρινήσεις σας και την πολιτική θέληση που δείχνετε να προχωρήσετε προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό επιθυμούμε και εμείς εδώ στην Ευρώπη. Ελπίζω δε Δεν είμαστε εμείς να εξετάσουμε τη δυνατότητα για την Ευρώπη να τηρήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο ασφαλώ ε, θα θελήσουν να συζητήσουν και κάποιοι συνάδελφοι. Έχουν ζητήσει το λόγο ήδη. Η κυρία Θεοχάρου πρώτη, παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. First of all... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη προ του διακεκριμένου και θαραλέου ε, ομιλητέ μα που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να φερθώ σε ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, ότι εδώ στην είσοδο της αίθουσα μας κάποιοι μοιράζουν αυτό το φυλάδιο, πράγμα το οποίο αντιβαίνει στον κανονισμό του Κοινοβουλίου και αποτελεί προσβολή για τον λαό της Κύπρου, την Κύπρο, το Κοινοβούλιο, τους βουλευτές που εκπροσωπούν εδώ την Δημοκρατία της Κύπρου. Εάν το γνωρίζετε, ποιο τους έδωσε την άδεια να το πράξουν. Η, πρόεδρο, η δεν έχω υπόψη μου τα έγγραφα αυτά, Όμω η Γραμματεία θα το εξετάσει αμέσω. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές να μας δώσουν πιο πολλές πληροφορίες για τις δίκες αυτές του Κατσεκά, του Κουρδικού Κογκρέσου. Ε, το φθινόπωρο που επισκέφθηκα την Τουρκία είχα την ευκαιρία να το θέμα αυτό μεταξύ άλλων. Και φαίνεται ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις συλλήψεων κάποιον ε, με την ε, κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, υποστήριξη προς τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή του κάθε συγκεκριμένα, χωρίς όμως ποτέ να είναι ε, οι αιτιολογίες ή κατηγορίες βάσιμες. Φερρυπίν κάποιος κατηγορήθηκε ε, γιατί το όνομά του εμφανιζόταν σε κάποιο CD με στοιχεία, που όμως τελικά ήταν μόνο το πρώτο όνομα και όχι το επώνυμο, κάποιος Αχμέτ Βερυπίν, ε, ή δεν βρέθηκε ποτέ ή δεν παρουσιάστηκε ποτέ το λόγο CD για να μελετηθεί και το καθεξής. Επίσης, από αυτά που άκουσα από συγγενείς ε, κρατουμένων, έχουν συλληφθεί και κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει καν πολιτική δράση, δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, δεν πέταξαν πέτρες και το Δηλαδή, ακόμα και αν θέλει κανείς μια τέτοια δραστηριότητα να την κατατάξει ως τρομοκρατική, Πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ή με τι άλλο, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν καν τέτοια δραστηριότητα. Ίσως παλαιότερα, αλλά σε ένα ούτως υπήν φυσιολογικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτές οι συλλήψεις είναι μάλλον τη χάρπαστας. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει πρόθεση να παταχθεί η τρομοκρατία, θα πρέπει να είναι πιο εστιασμένη η καταπολέμησή τη, όχι όποιον βρίσκουμε να συλλαμβάνουμε. Τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει εγώ, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω βέβαια την απόλυτη αλήθεια. Έχετε κι εσεί την εντύπωση ότι είναι κάπω ε, ε τυχαίε και τη χάρπα σε αυτέ τι συλλήψει. Και δεύτερον, για το ίδιο το Κουρδικό Κογκρέσο, το KCK. Πόσο πραγματικό θεωρείτε ότι είναι. Γιατί αυτό που ακούω επί το πλήστον είναι την, την κυβέρνηση να το κατηγορεί να λέει ότι υφίσταται, αποτελεί απειλή και τα λοιπά, συνιστά απειλή, αλλά τελικά να μην γνωρίζει κανείς τι ακριβώς πράττει. Εσείς θεωρείτε ότι υφίσταται, είναι κάτι το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υφίσταται. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα θέλω να, να ακούσω τις απόψεις. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και βεβαίως θα ξαναδώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Ε, τώρα η κυρία Λάτσφορτ, παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που έχετε οργανώσει. πέραν των πολύ σοβαρών ανησυχιών ως προς την κατάσταση στην ποινική δικαιοσύνη και την κατάχρηση θα έλεγα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας που όπως υπόθηκε μας έχει φέρει σε 9.000 υπόπτους σε προσωρινή κράτηση. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως πρώτα τον ε, κύριο Πρεσβευτή. το εξή. Εμείς περιμέναμε ότι ο Πρωθυπουργό θα συνέχισε μια πολιτική στρατηγική με στόχο την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Πράγμα το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται έχει βαλτώσει αν δεν έχει από ό,τι φαίνεται εγκαταλειφθεί τελείω. Υπάρχουν στη φυλακή από ό,τι γνωρίζω ε, βουλευτές τώρα, εκλεγμένοι βουλευτές του ΜΠΕΝΤΕΠΕ. Είχαν από ό,τι φαίνεται φυλακιστεί πριν από την ε, εκλογή τους ε, και έτσι τώρα δεν μπορούν να αποφυλεξτούν, αλλά αυτό ε, δείχνει ουσιαστικά τι παθαίνει κανείς όταν βρίσκεται στο λάθος μέρος. Βεβαίω, εγώ καταδικάζω περίφρασα την τρομοκρατία, την πραγματική τρομοκρατία, αλλά θα πρέπει να αναστήσουμε και μια λύση η οποία θα απαιτεί βέβαια δέσμευση και αποφάσει από την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα και την παρουσία ερετών εκπροσώπων των Κούρδων. Και από ό,τι έμαθα πρόσφατα έγινε επιδρομή τη αστυνομία και έρευνα στο σπίτι τη Λιλά Ζάνα. Αυτό δεν μα οδηγεί πουθενά βέβαια. Δεν μα προχωρεί προ μια λύση πολιτική του Κουρδικού. Μήπως τελικά δηλαδή κάνουμε ανάποδα κουπί. Και το άλλο, ως σχόλιο περισσότερο, γιατί δυστυχώς η Τουρκία δεν είναι η μόνη χώρα η οποία έχει ασαφή όρια μεταξύ των τρομοκρατικών ε, ε, εγκλημάτων και της ε, υπερβολικής χρήσης βίας η πατρίδα μου, γιατί και η Ευρώπη εν γέννη, αλλά ιδιαίτερα η πατρίδα μου για την οποία μπορώ να μιλάω, έχει πρώτη χαρακτηρίσει ως έγκλημα την ε, ε, υποστήριξη ε, της τρομοκρατίας, τους επένους προς την τρομοκρατία, πράγμα το οποίο φτάνει να αγγίζει ακόμη ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν με κάποια θετικά λόγια. Ε, και πρόσφατα ακούστηκε, ε, μάλλον ε, χαρακτηρίστηκε ως έγκλημα και η δημόσια πρόκληση τρομοκρατίας, έστω και αν αυτό δεν γίνεται με άμεσο τρόπο, αλλά απλώς αποτελεί κίνδυνο να διαπραχθούν τρομοκρατικές πράξεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι ο στόχος των οποίων εσφαλμένα ναι, επιδιώκει ο τρομοκράτης είναι ένας θεμητός στόχος, όχι το μέσον, αλλά κινδυνεύει να διωχθεί διότι φαίνεται σαν να ε, υποστηρίζει την τρομοκρατική δράση. Εδώ λοιπόν είναι πολύ ασαφή τα όρια και όσο περισσότερο ενισχύουμε αυτή την την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και όσο πιο πολύ καταπιέζουμε ή καταστέλουμε αυτές τις απόψεις αντί να προσπαθούμε να, ε, να εστιαστούμε σε εκείνους που ρητά υποθάλπουν ή ε, υποδαβλίζουν καλύτερα τρομοκρατικές πράξεις. Θα μπορούσαμε να δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Γιατί τελευταία ανάλυση πολλά είναι τα, τα δεινά που έχουμε δει το τελευταία, τα τελευταία δέκα χρόνια στο όνομα της τρομοκρατίας. Και στο θα μπορούσαμε να δώσουμε καλό παράδειγμα και στην Τουρκία εμείς με μια καλύτερη νομοθεσία πλευρά της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούτφορτ. Ας προσπαθήσουμε και οι δύο να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παράνομων συλλήψεων από την CIA, το πρόγραμμα της CIA. Εσύ και, εσείς και εγώ στον ίδιο αγώνα. Ο κύριος Μπάντλενερ ναι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά. Για την κυρία Λάτφορντ θα έλεγα δεν νομίζω ότι τέτοιου είδου μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν καταλαβαίνω για αυτά που λέτε γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για την Τουρκία και τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί. Δεν πρέπει να τα υποβαθμίζουμε όπως πράξετε εσείς. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω, νομίζω θα ήταν καλύτερο να κάνουμε αυτή την ακρόαση στην Τουρκία και να καλέσουμε τους εκπροσώπους της ε, τους εκπροσώπους αυτούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μιλήσουν και ενώπιον του τουρκικού κοινοβουλίου. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορούσατε να επαναλάβετε αυτές τις παρεμβάσεις στην Τουρκία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους Τούρκους βουλευτές της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη στιγμή που ήρθε στην εξουσία το κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Γιατί πώς Μπορεί η Τουρκία να συνεχίζει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμείς να συνεχίζουμε να συζητάμε με την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, όπως δεν έχει κάνει και τίποτα για την κατοχή της Κύπρου. Επανερχόμαστε στα ίδια θέματα και η Τουρκία εξακολουθεί το χαβά της. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσουμε και τη δική μας συμπεριφορά. Γιατί απλώς μιλάμε και τίποτα άλλο. Και το ίδιο αφορά το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας και την άρνηση αυτής της γενοκτονίας στην Τουρκία. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά είναι δυνατόν <clears throat> να είναι παράνομο να λέει κανείς ότι η Τουρκία δεν έκανε γενοκτονία. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, μάλλον να είναι παράνομο να λέει κανείς ότι η Τουρκία κάνει γενοκτονία, στην Τουρκία εννοεί ο μιλτής Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία, πρέπει να υπάρχουν δυνατότητα γελιογραφιών με τον προφήτη ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά τίποτα από αυτά δεν γίνονται στην Τουρκία. Επίσης έχουμε το πρόβλημα του ίντερνετ στην Τουρκία και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί τι έχει να πει ο κύριος Πρεσβευτής για το θέμα αυτό και πιστεύετε εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και πότε μπορεί να υπάρξει ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριε Μαντλέν, Μαντλενέρ. Είναι ένα νέο έτος το 2012 για να, μια μεγάλη ευκαιρία να έχετε μια μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερη ισορροπία στα λεγόμενά σας. Ο κύριος Κλούτε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές που είχαμε για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ξέρω και από την τουρκική πλευρά δεν είναι εύκολο να επικρίνει κανείς αυτή την κατάσταση και αναγνωρίζω πραγματικά τη συμβολή σας. Θέλω να ξεκινήσω με αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρεσβευτά. Πιστεύω, καταρχήν, ότι στην Τουρκία υπάρχει αυτή τη στιγμή <clears throat> μια σύγκρουση μεταξύ του κουρδικού τμήματος του πληθυσμού και των υπολείπων. Αυτό δεν έχει να κάνει με τρομοκρατία. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί με στρατιωτικά μέσα, μόνο με πολιτικές ενέργειες. Συμφωνώ με την κυρία Λούτφορτ ότι αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα που δεν μπορεί να επιληθεί με κατασταλτικά μέσα, με εφαρμογή του ποινικού κώδικος, με διώξεις ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ένοπλοι μαζί με το ΠΚΚ θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της λύση, όπως ακριβώς έγινε και με τη διαδικασία ειρήνευσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό, αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα της επίλυσης διαφορών και, της, και συγκρούσεων ξέρουν ότι μόνο με πολιτικό τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν αυτέ οι συγκρούσει. Θέλω λοιπόν να σα ενθαρρύνω να προχωρήσετε προ αυτή την κατεύθυνση. Ήδη πριν από δύο-τρία χρόνια υπήρξαν κάποιε προσπάθειες από την τουρκική κυβέρνηση, κάποια ανοίγματα και εγώ ήμουν ιδιαίτερα θετικό για τα θέματα αυτά, αλλά μετά από τι εκλογέ του περασμένου Ιουνίου έχουν ουσιαστικά σταματήσει αυτέ οι ενέργειε. θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορέσουν να προχωρήσουν και πάλι αυτέ οι προσπάθειε ανοίγματο και συμφιλίωσης. Κάτι ακόμα. Βλέπω επίσης ότι μεταξύ της ε, Τουρκίας και ορισμένων κρατών μελών υπάρχουν στενές επαφές που οδηγούν σε ορισμένες χώρες όπως τη δική μου χώρα να υπάρξει πίεση εναντίον των ε, κουρδικής καταγωγής ε, διαμενόντων από την Τουρκία που διαμένουν στις χώρες μας αυτές. Ε, ορισμένοι καλεσμένοι μου από το κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας, το 5 ε, υπέστησαν διάφορες ε, ταλαιπωρίες. Η κυρία Ζάνα που είχε έρθει στην ε, Γερμανία με την πίεση της ε, τουρκικής κυβέρνησης συνελήφθη. Επομένως δεν νομίζω ότι και εμείς φυλακή 40 Δεν νομίζω ότι αυτά είναι θετικά ούτε από την τουρκική πλευρά ούτε από τη γερμανική πλευρά. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να σταματήσει αυτή την ε, αντιμετώπιση η τουρκική κυβέρνηση γιατί με κανένα τρόπο δεν ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων και φυσικά δεν θεωρώ και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης ότι είναι επικοδομητική σε σχέση με τα θέματα αυτά. Πάλι ένα ερώτημα για τους τρεις ομιλητές μας. Πρόσφατα στη Δανία υπήρξε μια απόφαση για την τηλεόραση Rose που θεωρεί ότι που θέτει μεγάλη πίεση στη Rose TV ως, κουρδικού, ως κουρδικό κανάλι λέγεται ότι υπήρξε μια πίεση από το ΝΑΤΟ για να ληφθεί αυτή η απόφαση μετά από αίτηση της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να το αποδείξω, αλλά αυτό κυκλοφόρησε ως φήμη στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτή η απόφαση προεκλήθη πράγματι από μια πίεση της Τουρκίας. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα αυτό και πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις και επιπλέον να θέσω το ερώτημα αυτό στον κύριο Αταλάη. Έθεσε αυτό το ερώτημα, αναφέρθηκε σε αυτό προηγουμένως θα ήθελα να ξέρω από τη δική σας πλευρά τι θα ήταν χρήσιμο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ή κάτι διαφορετικό για να υποστηρίξουμε τις δικές σας προσπάθειες. <clears throat> Γιατί ο στόχος μας είναι η Τουρκία σαν υποψήφια χώρα να εκπληρεί όλα τα πολιτικά κριτήρια. Και επίσης η δημοκρατία θα πρέπει να υπάρχει και στην κρατική, στον κρατικό μηχανισμό και σε όλη την κοινωνία, αλλά όχι μονάχα σε ένα τυπικό επίπεδο, αλλά ενσωματωμένη σε μια πρακτική και σε καθημερινό επίπεδο. Θα ήθελα να ξέρω τι θα ήταν λοιπόν από τη δική σας πλευρά απαραίτητο για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την ε, θέση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα αν θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις ερωτήσεις μας. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Πρόεδρε, ε, η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δείχνει ε, πόσο σωστά επελέγει αυτό το θέμα συζήτησης και με αυτούς τους προσκεκλημένους και τον ε, κύριο Νισελ και τον κύριο Αταλάη και την ε, κυρία Σινκλέρ Βέμπ. Ε, που κάνανε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές παρεμβάσεις. Βεβαίως και ο, ο, πρέσβης της Τουρκίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνω ότι είχε μια πολύ καλή παρέμβαση. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ο κύριος Ινσέλ αναφέρθηκε και έκανε ένα σχόλιο και μια αξιολόγηση για την εξελισσόμενη δικαστική μεταρρύθμιση Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρέμβασή του, αλλά και τα τελικά του σχόλια. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί και για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άκουσα επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κύριο Αταλάη τα προβλήματα που έχει συναντήσει στην πορεία άσκησης της αποστολής του. Και εκεί ήθελα από αυτό έκυψε κάτι που, με, ε, που θέλω να αναδείξω. Βεβαίως η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι ένα ζήτημα. Όμως, από αυτά που είπε ο κύριος Σανταλάη, προκύπτει και μία κουλτούρα αυθαιρεσίας των αρχών. Αυτή η κουλτούρα αυθαιρεσίας δεν φαίνεται να μπορεί να λυθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις ή αναθεωρήσεις θεσμικές και εκεί αναδεικνύεται και ο ρόλος που έχει η αστυνομία. Η αστυνομία ως το πρώτο τμήμα της εξέλιξης μιας υπόθεσης. Και εκεί θα ήθελα να έχω την γνώμη τους πώς αξιολογούν την ποιότητα της, του έργου και το πώς ασκεί τα καθήκοντά της η αστυνομία και πόσο καλά συνεργάζεται ή τι θα πρέπει να γίνει για να συνεργάζεται καλύτερα με τη δικαστική εξουσία. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, φοβάμαι ότι δεν θα ακούσω την απάντηση γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση, αλλά είναι μια, συνεισφορά, μια προσπάθεια συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Merci, Obligé... Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Συγγνώμη που ήμουν αυστηρή. Η κυρία Σαλκέ. Σα Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία αυτής τη πολύ σημαντική συνεδρία. Δεν είμαι μέλος της JPC αλλά της Επιτροπής των Εξωτερικών και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερως για τα θέματα της Τουρκίας. Κύριε Πρεσβευτά, μιλήσατε για τις καλές προθέσεις, μιλήσατε για, την για τον ενεξελίξη εντατικό δημόσιο διάλογο. Εγώ έχω τα τελευταία τρία χρόνια ε, επισκεφτεί την Τουρκία τουλάχιστον 30 φορέ, πολλέ άλλε φορέ και πιο πριν ακόμη, αλλά μια και έχω το διαβατήριο το, το καινούριο τα τελευταία τρία χρόνια, μπορώ να μετρήσω μόνο αυτά. Ελπίζω ειλικρινά κάποια μέρα η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω πραγματικά ότι ο Τουρκικό λαό είναι πολύ ωραίο λαός, πολύ καλό λαός. Έχοντα λοιπόν ε, συνομιλήσει και με εκπροσώπου και τη κυβέρνηση αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου, διαπιστώνω ε, αισιοδοξία φιλοδοξία για την Τουρκία. Αλλά όταν μιλώ με άλλους ανθρώπους από την Τουρκία, διαπιστώνω δυσπιστία αντί των θεσμών, αυτολογοκρισία, ανησυχώ για, τους, ε, για την ομοθεσία για το ίντερνετ, ε, για την άσκηση, την, την ύπαρξη ελευθερίας του τύπου και ελευθερίας του διαδικτύου. Επαφές μου δε με πολλούς από τους επισήμους, της, ε, τους επισήμους φορείς ε, και την κυβέρνηση. Σαν απάντηση μου δίνουν μόνο την απόλυτη άρνηση των όσων ε, καταγγέλλονται εδώ. Αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει ότι έγινε μια προσπάθεια να καταστραφεί αδημοσίευτο βιβλίο. Και πιστεύω ότι αυτό που συζητούμε σήμερα περισσότερο απ' όλα είναι να κοιτάξουμε την ουσία, το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την πραγματική δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις ερωτήσεις. Εάν αναθεωρηθούν, να μεταρρυθμιστούν οι νόμοι, θα ισχύσει αυτή η μεταρρύθμιση και αναδρομικά. Δηλαδή μπορούν να ξανανοίξουν κάποιες υποθέσεις. Από πότε θα αρχίσει η ισχύ τους, των μεταρρυθμίσεων αυτών δηλαδή και η υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων, σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει αυτούς που βρίσκονται τώρα στη φυλακή. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει παρατηρητέ στι δικέ αυτέ μονίμως και όχι μόνο περιστασιακά. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμάτε το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητούμε έκθεση για την ε, διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας όπου μία από τις προτάσεις που περιέχει το κείμενο αυτό στο σχέδιό του αναφέρεται τώρα σε πιο στενή συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά εδώ υπάρχει σαφής αντίφαση ως προς την εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών, ε, του αντιτρομοκρατικού νόμου. Και επίσης, κάτι στο, το οποίο πιστεύω συμμερίζονται τόσο Ευρωπαίοι όσο και πολλοί Τούρκοι πολίτες, η συνεργασία υπό την σημαία του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχει στηθεί εδώ ε, καθόλου είναι ότι πολλοί από αυτούς που κρατούνται είτε, είτε εν αποστρατεία είτε εν ενεργεία ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας με, με το ΝΑΤΟ και σε πώς κρίνεται το γεγονός ότι τόσο υψηλ, τόσα πολλά και τόσο υψηλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μπορεί να κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί αυτό νομίζω ότι ανοίγει μεγάλη συζήτηση και αποτελεί σοβαρότατο λόγο ανησυχίας. Και επίσης Επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να εκφράσω την ευχή η Τουρκία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, να αντεπεξέλθει στα υπεσχημένα και να εκφράσω επίσης την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει την Τουρκία περισσότερο από τις δράσεις της και όχι από τις προθέσεις της. Και σε ελπίσουμε ότι αυτές οι δράσεις και οι πράξει θα είναι πραγματικά δημοκρατικέ ώστε να επικρατήσει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκε για την ομορφή σας αυτή η παρέμβαση, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Σταφ, η κυρία Θεοχάρου και η κυρία Κοπά, προτού γυρίσουμε στους ομιλητές μας. Κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους τρεις ομιλητές, γιατί όλα όσα ανάφερα σήμερα είναι πολύ γνωστά. Η έκθεση του Τόμας Χάμεμπερκ, αλλά και η για πολλά χρόνια διαδικασία παρακολούθησης Τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι ένα από τα θέματα που με απασχόλησαν και εμένα προσωπικά γιατί ήμουν μέλο στο Συμβουλίο τη Ευρώπη. Και ακούγοντα σήμερα και την εκπρόσωπο τη Διεθνή Αμνηστίας και τον κύριο καθηγητή αλλά και τον ε, δικηγόρο πραγματικά είναι αυτή η εικόνα που είχα στο μυαλό μου. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση η οποία για μας τους Θεούς είναι αδιανόητη. Ε, άκουσα τον κύριο Αχμέτιν Σελ να μιλά ότι η μεταρρύθμιση έχει καλές προθέσεις αλλά όχι γερές βάσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ ε, προβληματικό γιατί το να λέμε ότι γίνεται μια μεταρρύθμιση και να μην γίνεται στην ουσία μια ριζοσπαστική αλλαγή νοοτροπίας, μηχανισμών παραπέμπει σε εποχές σκοταδισμού όπως πολύ σωστά έχετε πει του 1990 και αλίμονον εάν ο αριθμός των 3.000 το 2008 αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει το 2012 σε τριπλάσιο αριθμό. Αυτό είναι μια κραυγή αγωνίας από έναν καθηγητή και πραγματικά με, έχει συγκλονίσει. Διότι εδώ θα έπρεπε ο κύριος Πρέσβης να μας πει τρόπους ώστε οι ακαδημαϊκοί τουλάχιστον να βρουν απαντήσεις πώς μπορούν να τεθούν γερές βάσεις σε αυτήν τη μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και αναμένω μια απάντηση από τον πρέσβη. Δεν αρκεί νομίζω μια επιτροπή εποπτείας των μεταρρυθμίσεων. Γιατί, γιατί γνωρίζουμε πως όταν ορίζεται μια επιτροπή η διαδικασία για να κινήσει τις μεταρρυθμίσεις είναι πολύ γραφειοκρατική όταν αφορά δημόσιο τομέα. Και αν θα πάρει άλλα τόσα χρόνια για να υλοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις προς Θεού στο μεσοδιάστημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι προφυλακισμένοι ή είναι καταδικασμένοι μπορεί να χάσουν τις ζωέ του. Και εγώ έχω τη φιλοσοφία αλήθεια ότι όταν η δικαιοσύνη δεν απονέμεται έγκαιρα και όταν καθυστερεί ουσιαστικά δεν είναι δικαιοσύνη. Επομένω, το πρώτο ερώτημα μου είναι πώ να τεθούν γερέ βάσει σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει, κύριε Πρέσβη. Αναφέρομαι τώρα στον κύριο Ακίνα Ταλάη, ο οποίο έχει πει ότι αδυνατεί να εκτελέσει το έργο του. Ουέ και αλλήμον Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν μία δίκαιη λύση, όταν αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται και τα στοιχεία ακριβώς μαζεύονται ενώ είναι κρατούμενοι χωρίς να υπάρχει στοιχειώδες ένταλμα ε, σύλληψης. Για μένα είναι αδιανόητο να μπαίνουν στη φυλακή άνθρωποι χωρίς στοιχεία και όταν είναι φυλακισμένοι να μαζεύονται αυτά τα στοιχεία. Και εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Και το τρίτο ερώτημα αφορά την κυρία Έμμα Σικλέρ, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι ασχολείται με το θέμα της διεθνούς αμνηστίας. Τελειώνω, τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Έχω υπόψη μου την περίπτωση του κυρίου Ραγίπ Ζαράκολου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Τούρκων ε, της Ένωσης Publishers Union Committee ο συγκεκριμένος ε, έχει συλληφθεί γιατί ακριβώς είχε να δημοσίευτα ε, βιβλία και αρκετά από τα βιβλία που είχε ε, δημοσιεύσει αφορούσαν την αρμενική γενοκτονία. Η ερώτηση μου είναι πόσους ακόμα τέτοιους ανθρώπους, είτε συγγραφείς, είτε ακτιβιστές, είτε άλλους που έχουν συλληφθεί θα δούμε να βρίσκονται στις φυλακές και να μην βλέπουμε πραγματικά έναν τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση να πατάξει την κρατική τρομοκρατία που ασκείται. Ευχαριστώ. Okay, okay. Merci, merci beaucoup, monsieur. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταφ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λόγω ακριβώς της σοβαρότητας της κατάστασης στην Τουρκία, νομίζω ότι θα πρέπει να εκφραστούμε θετικά για το πακέτο το οποίο η κυβέρνηση έχει καταθέσει. Είναι η πρώτη, θα έλεγα, σοβαρή, συνολική προσπάθεια μεταρρύθμισης του δευτερογενούς δικαίου, ιδιαίτερα στα πλαίσια του ποινικού. Ελπίζω ότι ο ενθουσιασμός για τις μεταρρυθμίσεις, ο οποίος προέρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να χαρακτηρίζει και την υπόλοιπη κυβέρνηση, ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών. Το ερώτημά μου τώρα. Το βασικό σημείο εδώ είναι ο καταστατικός χάρτης και όχι το δευτερογενές δίκαιο. Uh, Δεν είναι το πρόβλημα στο παράγωγο τόσο δίκαιο όσο στο σύνταγμα της χώρας. Εμπνέει καταστάσεις και νοοτροπίες οι οποίες στην ουσία οδηγούν στο να στο ότι οι δυνάμεις ασφαλείας και οι δυνάμεις καταστολής και η δικαιοσύνη δίνει την εντύπωση ότι προστατεύει το κράτος πρώτα και τους πολίτες μετά. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα οι προσκεκλημένοι μας να μας πούν πώς θα υπάρξει μια κάποια αλληλοεπίδραση ανάμεσα στη μεταρρύθμιση του παραγόγου δικαίου ή του δευτερογενούς δικαίου και στην απαραίτητη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης. Θα υπάρξει μια παράλληλη διαδικασία οι προσπάθειες και από τις δύο κατευθύνσεις ε, θα προχωρήσουν με τρόπο συμβατό ή θα υπάρξει ένας χρονισμός ο οποίος θα επιτρέψει να προχωρήσει ο ένας κλάδος και να ακολουθήσει ο άλλος σε μια άλλη φάση. Λοιπόν, η αναφορά σας ε, ήταν για το νέο σύνταγμα προφανώς, η κυρία Θεοχάρους. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου στους ομιλητές, καθώς επίσης και σε όλους τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παλεύουν μέσα στην Τουρκία, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι οι πράξεις μέσα σε ένα χώρο που έχει αυτά τα δεδομένα, όπως μας τα έχετε περιγράψει, μετράνε χίλιες φορές περισσότερο από πράξεις που γίνονται σε ένα χώρο σαν αυτόν εδώ πέρα όπου μπορούμε ελεύθερα να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ό,τι θέλουμε, ειδικά όταν αγωνίζεστε για να υπερασπιστείτε κάποιους ανθρώπους. Και ελπίζω ποτέ να μην ακουστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξανά εκείνο που ακούσαμε αρκετά φορές να λένε ότι ναι είναι κακή η κατάσταση αλλά ξέρετε επειδή όγκος συναλλαγών της Τουρκίας, η οικονομία και όλα αυτά τα ζητήματα είναι συντριπτικά πάρα πολύ ισχυρά, τότε μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την ιστορία. Είναι ζωτική σημασία. Εκφράζω τον θαυμασμό μου σε όλους τους αγωνιστές που προσπαθούν να κάνουν πιο καλή, πιο δίκαιη την, την τουρκική κοινωνία και το δίκαιο. Τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω τις έχουν ήδη πει οι συνάδελφοι. Αντιλαμβάνομαι ότι μας πιέζει και ο χρόνος. Απλά μια ερώτηση ίσως είναι άσχετη, γι' αυτό μη μου την απαντήσετε αν δεν σας ε, αν δεν την κρίνετε ότι εντάσσεται σε αυτά που θέλετε να μας πείτε, γίνεται χρήση χημικών όπλων εναντίον του κουρδικού πληθυσμού ή όχι. Ευχαριστώ. Κυρία Κοπά, ακούσαμε σήμερα εξαιρετικές εισηγήσει για τις αδυναμίες του νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο αντιτρομοκρατικός νόμος άρα η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επιβάλλεται άμεσα και είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, το δικό μου πολύ σύντομο σχόλιο αφορά όμως στην ουσία του προβλήματος. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος βρέθηκε για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά α, κινήσεις, προβλήματα που, ε, που δημιουργούνται μεταξύ Τούρκων πολιτών κουρδικής καταγωγής. Το πρόβλημα λοιπόν στην ουσία είναι το κουρδικό πρόβλημα ό,τι νομοθετική ρύθμιση και αν υπάρξει ό,τι αλλαγή του νομικού πλαισίου ακόμα και κατάργηση πλήρης του αντιτρομοκρατικού νόμου δεν μπορεί να υπάρξει ε, πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν δεν λυθεί το ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα που είναι το κουρδικό πρόβλημα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην τουρκία δεν βλέπουμε καμία κίνηση προς την κατεύθυνση της επίλυσης του. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κοπά. Ξαναγυρίζουμε γυρίζουμε στους προσκεκλημένους Ο κύριος Πρέσβης, ο οποίος ε, είναι το αντικείμενο πολλών ερωτήσεων, εάν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά ως Τούρκος πολίτης. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πού βρισκόμαστε. Το κουρδικό θέμα. Πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε καν να προφέρουμε τη λέξη Κούρδος. Τώρα έχουμε ένα κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος εκπέμπει στα κουρδικά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Εμείς διαχωρίζουμε το θέμα της τρομοκρατίας από το κουρδικό. Οι τρομοκράτες δεν ξέρουν ποιοι είναι. Αλλά το κουρδικό θέμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η ελπίδα μας είναι ότι όταν έχουμε το νέο σύνταγμα, το οποίο είναι υποσυζήτηση, όταν έχουμε ένα νέο σύνταγμα, ένα πολιτικό σύνταγμα, όχι στρατιωτικό, θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα. Για το σχέδιο νόμου τώρα που ανέφερα, θα πρέπει να διευκρινίσω μερικά θέματα, γιατί ίσω υπήρχαν κάποιες ελλείψεις αυτά που είπαμε προηγουμένω. Πρώτα απ' όλα αυτό ο νόμο θα υποστηρίξει την ελευθερία έκφραση. Αν υπάρχουν προβλήματα λοιπόν τώρα, τα προβλήματα αυτά δεν θα υπάρχουν μετά από την εφαρμογή αυτού του νόμου. Ρωτήσατε πόσο καιρό θα χρειαστεί αυτή η διαδικασία. Μάλλον δύο μήνες το maximum στο κοινοβούλιο μας. Η ομάδα παρακολούθησης για τα θέματα αυτά αποτελείται από βουλευτές και από μέλη του κρατικού μηχανισμού και εγώ παρακολουθώ αυτές τις συζητήσεις και υπάρχει μια πολύ έντονη και ζωντανή συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει. Η νομοθεσία αυτή δεν θα είναι απόλυτα αναδρομική αλλά θα αντιμετωπίσει πολλά ε, θέματα που είναι ακόμα ανοιχτά. Πολλού φακέλους που είναι ακόμα ανοιχτοί. Ναι, επομένως έχει κάποιο, ένα αναδρομικό χαρακτήρα. Μπορείτε εσείς επίσης να είστε παρόντες στις ε, δίκες. Για τα χημικά όπλα, όχι βέβαια, αυτό είναι κάτι το φοβερό που λέτε. Και επίσης για αυτό το οποίο είπε ο διακεκριμένος ε, βουλευτή. Εγώ άκουσα δύο λέξεις η επιδείνωση και η δικτατορία. Ίσως μιλάτε για μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τουρκία, αλλά μπορείτε να έρθετε στην Τουρκία, πείτε ό,τι θέλετε και θα δείτε ότι δεν είναι η Τουρκία την οποία εσείς νομίζετε ότι έχετε ενώπιον σα. Σας ευχαριστώ για τι συγκεκριμένε σας απαντήσει. Κύριε Ινσέλ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί, στις περισσότερες από αυτές τουλάχιστον. Να κάνω εδώ μία διευκρίνηση. Πολλοί που πήραν το λόγο, όπως και ο κύριος Πρέσβης, είπαν ότι από τη μία υπάρχει το θέμα του νόμου και από την άλλη η ερμηνεία και η εφαρμογή του νόμου από πλευράς του δικαστικού προσωπικού και από πλευράς επίσης και των δυνάμεων καταστολής. Είναι αλήθεια ότι στην Τουρκία υπάρχουν κάποιες νοοτροπίες, θα έλεγα αυταρχικές, οι οποίες ε, ε, πραγματικά χαρακτηρίζουν πολλές φορές τις συμπεριφορές των δικαστικών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, κάποια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επιληθεί υπό κανονικέ συνθήκες χωρίς τη χρήση βία, πάρα πολύ συχνά ξεφεύγει από τον έλεγχο και οδηγούμεθα στη χρήση βία. Υπάρχει και κάτι το διαφορετικό εδώ. Ο δικαστικός κόσμος θα έλεγα, ιδιαίτερα στον ποινικό τομέα, είναι πάρα πολύ στραμμένος προς το κράτος προς την προάσπιση των κρατικών συμφερόντων. Γίνεται μια προσπάθεια, είναι σαφές από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και σε επίπεδο του δικαστικού προσωπικού που θα πρέπει να εμπνέεται περισσότερο από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά παρόλα αυτά κάποια ρεφλέξ αυταρχικά εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο αναφερθήκατε πολλοί από εσάς η κυβέρνηση, τουλάχιστον κάποια μέλη της κυβέρνησης σε βάση περιπτώσει, δεν είναι θα έλεγα εκτός ευθυνών σχετικά με τα μηνύματα τα οποία σαν κυβέρνηση αποστέλουν προς τους δικαστές και προς τις αστυνομικές αρχές σχετικά με την καταχρηστική χρήση από πλευρά ορισμένων αρχών, από πλευρά δικαιοσύνη. Εδώ και ένα μήνα, σαν παράδειγμα, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, μετά από τι κριτικέ τι οποίε ακούσαμε και μοιάζουν με αυτά που ακούσαμε πριν, ο Υπουργό Εσωτερικών, ε, ναι, Εσωτερικών, είπε σε μία συνάντηση των ομαρχιακών αρχών, σε μία συνάντηση εργασία στην Κεντρική Ανατολία, ότι θα μπορούσαμε να συμμετέχει κανείς σε τρομοκρατικές ενέργειες και να διαπράττει τρομοκρατικά εγκλήματα, όχι μόνο χρησιμοποιώντας όπλα, αλλά <clears throat> και ασκώντας δημοσιογραφικές δραστηριότητες, λογοτεχνικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργό ότι μπορεί κανείς να προωθήσει, να διασπείρει τρομοκρατικές ιδέες μέσω τη δράσης του ως δημοσιογράφου, καλλιτέχνη, ποιητή κτλ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι ο υπουργό με ένα πολύ, ε, θα έλεγα, καταχρηστικό τρόπο διευρύνει την ερμηνεία των τρομοκρατικών ενεργειών και όταν βλέπουμε τον Υπουργό Εσωτερικών να έχει μια τέτοια σκέψη καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολο οι αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμόζουν την ίδια λογική. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Δεν λέω ότι το σύνολο των μελών της κυβέρνησης αντίστοιχα μηνύματα εκπέμπουν. Όχι, υπάρχουν άλλα μέλη της κυβέρνησης ένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, σαν παράδειγμα πριν μερικούς μήνες, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εκ νέου ορισμός της τρομοκρατικής δράσης και να γίνει μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης από τη μία, την ελευθερία διαδήλωσης από την άλλη και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, ο υπουργό Εσωτερικών είναι, ε, επηρεάζει πολύ περισσότερο την αστυνομία από ότι ο άλλος Υπουργός. Ένα δεύτερο παράδειγμα πρέπει να σας δώσω. Δυστυχώς μετά από τη σύλληψη του Σενέρ και του ΣΥΚ, ο Πρωθυπουργό μας είπε κάτι το οποίο χαρακτηρίζω ατυχές. Είπε ότι ένα βιβλίο πολλές φορές είναι πολύ πιο επικίνδυνο από μία βόμβα. Ε, ίσως σε ιδεολογικό επίπεδο κάτι τέτοιο να ισχύει. Αλλά μία βόμβα είναι μια βόμβα και ένα βιβλίο είναι ένα βιβλίο. Και να κάνει κανείς μια τέτοια σύγκριση, μια τέτοια αναλογία, στην ουσία διευρύνει ερμηνεύοντας την τρομοκρατική δράση. Και γι' αυτό λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνωρίζουμε ότι κάνει μια πιο συστηματική προσπάθεια. Τώρα ε, υπάρχει ο καλός και ο κακός στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλει να παίξουν. Ίσως δεν είναι όμως ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς θέλουμε μήνυματα να εκπέμπονται θετικά προς την αστυνομία και τη δικαιοσύνη για να βοηθήσουν την κατάσταση. Τέλος, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος χώρος υπερβολικό βάρος στις ανακριτικές υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται από πλευρά της ε, ειδική αστυνομίας. Παρά τις ε, υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία, παρά τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Τουρκία δεν έχουμε δικαστική αστυνομία. Έτσι λοιπόν, το δικαστικό σώμα δεν έχει στη διάθεσή του μια αστυνομική δύναμη ανεξάρτητη, σε άμεση σχέση με την εισαγγελία και έτσι η αστυνομία έχει πλήρη ελευθερία να κάνει όλες τις ανακρίσεις και γι' αυτό ακριβώς και αυτό το γνωρίζει ο Αταλάη καλύτερα από μένα ο φάκελος ενημέρωσης που προέρχεται από την αστυνομία σε μία πρώτη φάση μετά από ένα συμβάν φτάνει στον εισαγγελέα και αυτόματα ο φάκελος αυτός μετατρέπεται σε κατηγορητήριο το οποίο είναι διευρυμένο εκ των προτέρων από πλευράς ε, του εισαγγελέως ε, εις βάρος ε, του κατηγορουμένου. Λοιπόν, ο φάκελος αυτός δεν εγκαταλείπει ποτέ ο αστυνομικός, ο ανακριτικός τον φάκελο του, ε, κατηγορουμένου. Και μέχρι ακόμα και το ανώτατο δικαστήριο υπάρχουν πάντα στοιχεία του πρώτου φακέλου που συνέταξε και συνέφεσε η αστυνομική ανακριτική αρχή. Τίθεται ένα θέμα λοιπόν εδώ ισορροπία των δυνάμεων και βάρους υπερβολικού του ρόλου της αστυνομίας σε σχέση με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα στα θέματα τα ποινικά ή τα υποτιθέμενα ποινικά. Είναι αλήθεια ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις. Θα σας, θα σας στεναχωρήσω. Η Τουρκία δεν είναι δικτατορία. Είναι μια χώρα όπου υπάρχει θάρρος, υπάρχει κριτική, υπάρχει πολιτική σκέψη, πολλοί ασκούν την κριτική αυτή, υπάρχουν πολλές ενώσεις, πολλοί σύλλογοι, κάνουν ελεύθερες συνεδριάσεις όπως και οι δικηγορικοί σύλλογοι κτλ. Έχουν υπάρξει όμως βελτιώσεις. Έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, και όπως είπα υπάρχουν βελτιώσεις και σε άλλους τομείς όπως τα βασανιστήρια στους αστυνομικούς σταθμούς. Δεν έχουν εξαφανιστεί φυσικά κατά 100% αλλά έχουν μειωθεί κατά πολύ και τώρα η αστυνομία δεν βασανίζει για να ομολογήσει ο κατηγορούμενος. Έχουν πιο τεχνικά αναπτυγμένα μέσα, δεν έχουν ανάγκη εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούν νόμιμα ή παράνομα τις επικοινωνίες, εν πάση περιπτώσει ο, ο ίδιος ο κατηγορούμενος ε, ανακαλύπτει αυτό το οποίο είχε πει αυτό το οποίο ήθελε να πει και πολλές φορές ο κατηγορούμενος βλέπει ότι η αστυνομία ξέρει πιο πολλά από αυτόν από ότι ο ίδιος για τον εαυτό του. Η αστυνομία λοιπόν δεν βασανίζει πλέον. Τώρα, αν έχει υπάρξει μια ουσιαστική βελτίωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Ζαρακόλ από ό,τι γνωρίζω δεν φυλακίστηκε γιατί δημοσίευσε βιβλία, αλλά γιατί δούλεψε προς αναγνώριση της γενοκτονίας. Δεν γνωρίζουμε όμως εμείς και ούτε αυτός γνωρίζει γιατί έχει συλληφθεί. Περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν ποιο είναι το κατηγορητήριο στην περίπτωση του κυρίου Ζαρακόλ. Εξάλλου υπάρχει και ένας πολιτισμός θα έλεγα αυθαιρεσίας στην Τουρκία. Αυτό είναι κάτι το οποίο βαρύνει ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα. Σας είπα ότι έγιναν πολύ σημαντικές συναντήσεις οι οποίες άσκησαν ουσιαστική κριτική στην κοινοβουλευτική και στην κυβερνητική δράση χωρίς να κατηγορηθούμε. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πολιτική η οποία μερικές φορές μπορεί να γίνει κατασταλτική και αυτό ανεξέλεγκτα. Αυτό λοιπόν που είναι προβληματικό σήμερα είναι οι ήχοι που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Οι ψήθυροι που προέρχονται πολλές φορές από αστυνομικές αρχές ή από κάποιες ομάδες που δεν γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις οποίους αυτές, αυτούς ψιθύρους υπάρχουν, ε, θα έλεγα, θα υπάρξουν μάλλον κύματα συλλήψεων, διανοουμένων κτλ και μία φορά στις δύο γίνεται αυτό. Αυτές οι συλλήψεις πολλές φορές γνωστοποιούνται αν θέλετε πριν τελεσθούν και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Ένα κλίμα στα πλαίσια του οποίου η αφαιρεσία σοβεί. Έχουμε λοιπόν μία Τουρκία από τη μία των ελευθεριών και έτσι εγώ και ο συνάδελφος Αταλάη δουλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να μας ενοχλεί κανείς, εμένα δεν με ενοχλεί κανείς, αλλά το ίδιο που κάνει κάποιος άλλος δυστυχώς οδηγεί στην παρενόχλησή του. Υπάρχει μια πλήρης αυθαιρεσία σε σχέση με τον καθορισμό των ορίων της νομιμότητας και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα το οποίο τίθεται σήμερα στην Τουρκία. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια χώρα φυλακή, όχι, πόσο μάλλον υπάρχουν χώροι ελευθερίας αλλά η χώρη αυτή ελευθερίας και το πέρασμα ανάμεσα στον χώρο ελευθερίας και την καταστολή είναι πάρα πολύ σκοτεινό και θολό και τόσο θολό έτσι ώστε να μην μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία είναι μια απόλυτα δημοκρατική χώρα. Τώρα, η το Σύνταγμα προκαλεί τα προβλήματα αυτά. Ναι, πράγματι αυτό γίνεται. Το Σύνταγμα έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 1982. Άνω του 50% των άρθρων έχουν τροποποιηθεί. Αλλά το Σύνταγμα το οποίο προετοίμασαν οι στρατιωτικοί και οι αυταρχικές πολιτικές προσωπικότητες μετά το πραξικόπημα στη δεκαετία του 80 οδήγησαν σε ένα σύνταγμα του οποίου η καρδιά πιέζει την, την εξουσία να λειτουργήσει με αυθαιρεσία. Πρόκειται για ένα σύνταγμα του οποίου η διάρθρωση είναι μια διάρθρωση που οδηγεί στην αυθαιρεσία, οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση, οδηγεί στον αυταρχισμό σε μια προσπάθεια υπεράσπισης του κράτους εις βάρος της κοινωνίας. Οπότε πρέπει να πει κανείς ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα πριν να αλλάξουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πιστεύουν όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα από, τότε, από το 1992 και μετά. Αλλά από το 1992 και μετά το Σύνταγμα δεν το έχουμε αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια δυνατότητα εδώ Υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνταγματικής μεταρρύθμισης υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν θα καταλήξουμε γρήγορα από ό,τι φαίνεται και αν θέλουμε να υπάρξει συζήτηση στα πλαίσια αυτών των αρχών δεν θα περιμένουμε να επιτελεστούν. Οι συζητήσεις αυτές απαιτούν οι αφαιρεσίες όπως οι απαράδεκτες προφυλακίσεις, οι απειλές που δημιουργούνται και που οδηγούν σε αυτολογοκρισίες. Όλες αυτές οι απαράδεκτες καταστάσεις πρέπει να σταματήσουν. Περιμένοντας λοιπόν τις συνταγματικές αλλαγέ. Οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε ήδη σημειώσει στο, ε, στο κείμενο που προετοιμάσαμε θα πρέπει να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να περάσουμε σε μια συνταγματική αλλαγή στα πλαίσια μιας ισχυρής δημοκρατίας, μιας αντιπροσεπευτικής δημοκρατίας, μιας πιο τακτοποιημένης αν θέλετε δημοκρατικής τάξης. Λοιπόν, υπάρχει ένα στενό, ένα στενό επίσης, ένα στενό σύνδεσμος ανάμεσα στα δημοκρατικά θέματα στην Τουρκία και στο κουρδικό. Η κατάσταση στα πλαίσια του κουρδικού δημιουργεί μια μόνιμη ένταση και από πλευρά της κυβέρνησης δυστυχώς υπάρχει ένας διαχωρισμός ιδιαίτερα τονισμένος, ιδιαίτερα ριζικός, απόλυτος θα έλεγα, ανάμεσα στο κουρδικό από τη μία και τους άμεσα εκλεγμένους εκπροσώπους από τους πολίτες της Τουρκίας, τους εκπροσώπους, τους κοινοβουλευτικούς δηλαδή, οι οποίοι ε, εμφανίζονται σαν εκφραστές του Κουρδικού από πλευράς του BDP. Η κατάσταση αυτή, αν θέλετε, προκαλεί καταχρήσεις, προκαλεί χρήση στην εφαρμογή των τρομοκρατικών ή αντιτρομοκρατικών καλύτερα διατάξεων γιατί η αστυνομία και το κράτος θεωρούν ότι ακριβώς η κυβέρνηση, το κράτος διαπιστώνουν μία θεμητή αν θέλετε αντίθεση και αυτό το κάνουν και τα εθνικιστικά κόμματα θεωρούν ότι υπάρχει μία αντιπολίτευση νόμιμη και μία αντιπολίτευση παράνομη, η οποία απειλεί την ασφάλεια της χώρας. Αυτό το πνεύμα, σύμφωνα με το οποίο ένα ανώμημα εκλεγμένο κόμμα, αναγνωρισμένο κόμμα, αποτελεί μη νόμιμη μορφή αντιπολίτευσης, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα και για το κουρδικό και για την αριστερή και ακροαριστερή αντιπολίτευση και για αυτούς οι οποίοι θεωρούνται από πλευράς της, ε, των ε, αρχών ασφαλείας επικίνδυνη για την δημόσια ασφάλεια, για την κρατική ασφάλεια και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις το είδαμε αυτό μετά από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδίδονται, απο, ε, μάλλον τους αποδίδουν ενέργειες βλαβερές για την κυβέρνηση, επικίνδυνες για την κυβέρνηση το ότι μπορεί οι διαδηλώσεις αυτές να θεωρούνται επικίνδυνες για την κυβέρνηση επειδή προέρχονται από μία συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία λογική, με μία νοοτροπία κατασταλτική και αντιδημοκρατική. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Καταρχάς παρακολουθώντας από κοντά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία και πράγματι συμβαίνουν πάρα πολλά στην Τουρκία και καλά και άσχημα. Θα πρέπει να μας υποστηρίξετε, να υποστηρίξετε αυτά τα οποία γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν η μεταρρύθμιση εν μέρη πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να την υποστηρίξουμε και να την υποστηρίξετε κι εσείς. Πρέπει να μας βοηθήσετε παράλληλα πιέζοντας την κυβέρνηση εφόσον έχετε την δυνατότητα ή να βοηθήσετε ακόμα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τα πολιτικά κόμματα με τα οποία σχετίζεστε μέσω των κοινοβουλευτικών αυτών επαφών έτσι ώστε τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα το κόμμα το οποίο βρίσκεται στην εξουσία και το οποίο είναι κατεξοχήν υπεύθυνο να είναι ευαίσθητο το κυβερνητικό αυτό κόμμα στην αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο κανόνων και όχι σε επίπεδο συγκυρίας. Θα πρέπει στην Τουρκία να ακολουθήσουμε μία μορφή αντιμετώπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι απλά πραγματιστική, αλλά μία διαδικασία διακανονιστική βασισμένη στο δίκαιο. Ευχαριστώ θερμά κύριε Αχμέτιν Σελ. Ήταν πολύ σαφή όλα αυτά. μα συνάρπασαν όλου και βέβαια σημαίνουν πολλή δουλειά και κινητοποίηση και από την πλευρά μα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα αίτημα παραδείγματι και καλό τους συναδέλφους να στηρίξουν την πρόταση σε μία ε, στην προσεχή συνεδρίαση το αίτημα για άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 των διαπραγματεύσεων που θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερε πιέσει προ την κυβέρνηση. Αυτά αφορούν βέβαια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα μπορούσαμε έτσι να πιέσουμε την κυβέρνηση για να προχωρήσει αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Και επίση πιστεύω ότι με την ad hoc ε, αντιπροσωπή ο κύριο Καρύμ που ήταν μαζί μα νωρίτερα αλλά δεν μπόρεσα να τον ε, παρουσιάσω στην Ομίγυρη ασχολείται λοιπόν με την υπόθεση αυτή των ε, δικών των δημοσιογράφων και έχει κάνει δουλειά που είμαι βεβαία θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για τους στόχους που περιγράψατε. Πριν ζητήσω να συμπληρώσει πολύ σύντομα ο κύριος Αταλάη την παρέμβαση του κυρίου Σέλ, θα ζητήσω από τους διερμηνείς μερικά ακόμη λεπτά. Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει, υπάρχει μια ανάγκη οι ομάδες που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμμετάσχουν στις προσπάθειες μεταρρύθμισης που γίνονται. Είναι απαραίτητο να πάρουμε στα σοβαρά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και να προσπαθήσουμε να τις επηρεάσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται ένας πραγματικός διάλογος με την τουρκική κυβέρνηση για τα σχέδια αυτά μεταρρύθμισης. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να προωθήσουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Και <clears throat> το γεγονός ότι πράττουμε κάτι τέτοιο, αυτό δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε τον, τις κριτικές μας, ότι αυτοφημονόμαστε και πάβουμε να ε, διαμαρτυρόμαστε για ορισμένα πράγματα. Θα πρέπει παρόλα αυτά να συμμετάσχουμε χωρίς να πάψουμε να επικρίνουμε, όχι με έναν τρόπο ο οποίος είναι αυθαίρετος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθύνσεις που έχει δώσει το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Νομίζουμε ότι αυτός είναι σωστός οδικός χώρο, ε, χάρτης. Αυτός είναι λοιπόν ο, αυτή είναι η αποστολή μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση. Αυτό πρέπει να είναι ένα κεντρικό κομμάτι της εργασίας μας πρέπει να υπάρξει πολύ καλύτερη διάκριση μεταξύ της ε, θεμητής έκφρασης απόψεων και της τρομοκρατίας στην Τουρκία. Δεν είναι θέμα μοναχα των ποινών ή τροποποίησης ορισμένων διαδικαστηριών. Δεν είναι θέμα αναστολής ή αναβολής της έκτησης ποινών. Θα πρέπει να πούμε στον πυρήνα του προβλήματος σε σαφείς ορισμούς και σε σαφή κριτήρια τα οποία θα καθοδηγούν τις ε, αποφάσεις των δικαστηρίων και την ομολογία του μέλλοντος. Και αυτό πρέπει να γίνει με υποστήριξη της κυβέρνησης. Για, την, για το KCK, κατσεκά, ε, υπάρχουν πράγματι πολλά προβλήματα με τη δικαστική εξουσία. Φαίνεται ότι ξεκινάνε όλα από τις ιδιαίτερες εξουσίες που έχει η αστυνομία, φτάνουν στα δικαστήρια, υπάρχει η παράταση της ε, προφυλάξης, υπάρχουν πάρα πολλά προβληματικά στοιχεία που είναι προβληματικά, ένας τεράστιος αριθμός και φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα της ίδιας νομοθεσίας. <clears throat> ναι. Πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα της υπεράσπισης στις δίκες δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι τα... Για το άτομο που αναφέρθηκε δεν ξέρουμε ακόμα τον κύριο Καλακόλ, δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα, ποιο ακόμα θα είναι το κατηγορητήριο, οπότε δεν μπορούμε ακόμα να αποφαθούμε. Εντάξει, αυτά είναι συντομία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σανκλέρ. Ο τελικός λόγος τον κύριο Αταλάη. Ε, ε, μια και δεν έχω πολύ χρόνο, θα συμπληρώσω πολύ σύντομα τα τελευταία, ό,τι δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα, μέσα σε δύο λεπτά μόνο. Πρώτον, ο ρόλος που θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να συμβάλλει δηλαδή στην υπόθεσή μας. Θα σα πω το εξή. Σήμερα παρουσιάστηκε στην Βουλή μία πρόταση μεταρρυθμίσεων στην ε, Τουρκία που είναι ανεπαρκής, που θα πρέπει να προχωρήσει με πολύ περισσότερα στοιχεία. Σε αυτό λοιπόν, στην προσπάθεια να εμπλουτιστεί αυτή η διαδικασία, μπορείτε να συνεργαστείτε με το τουρκικό κοινοβούλιο, αυτό το πιστεύω κράδαντα. Και μέσα από όλα τα κόμματα, με ανοιχτή συζήτηση, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει αυτή η προσπάθεια. Δεύτερον, ιδιαίτερα και πάνω απ' όλα, πριν από όλα τα επιμέρους θέματα, το ζήτημα που έχει μετατραπεί σε ανοιχτή πληγή στην Τουρκία, δηλαδή το ζήτημα της ε, ελευθερίας της έκφρασης που καταγράφεται, καταγγέλλεται ως τρομοκρατική πράξη και η διάρκεια λόγω της, ε, του κατηγορητηρίου της τρομοκρατίας της ε, προσωρινής κράτησης που είναι υπερβολική και η οποία ουσιαστικά εγγράφεται μέσα στη γενικότερη ε, δέσμη που ονομάζεται κράτος δικαίου και δίκαιη δίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ήρθε η στιγμή για πολύ θερμές ευχαριστίες. Ήταν πλουσία η συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα, συναρπαστική. Μας άνοιξε πολλούς δρόμους για διερεύνηση. Η προσεχή μας ε, μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τη συνεδρίασή τη που θα ασχοληθεί και με τη μεταρρύθμιση του συντάγματο και με την δικαστική μεταρρύθμιση και θα συναντήσει βέβαια και τον Υπουργό Εργίν της Δικαιοσύνης. Πιστεύω θα έχει πολλά να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μας έχετε ε, ανοίξει νέους δρόμους. Ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά, κυρία Αταλάη, κυρία Μασενκλέρ, κυρία Αχμέτιν Σέλ. Ευχαριστώ όλους αγαπητοί φίλοι.